Good morning, ladies and gentlemen. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρακαλώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Αθρώα η προσέλευση. Χθες ήμασταν πολύ πιο λίγοι, σήμερα είναι εντυπωσιακή η παρουσία σας. Ξεκινάμε με τις ψηφοφορίες και πρώτα με τη γνωμοδότηση της κυρίας Κωνσταντσε Κρέλ με θέμα τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στο Γενικό Προϋπολογισμό της Ένωσης. Ήταν χρονοβόρα η διαδικασία εκπόνησης της γνωμοδότησης, πλειάδα οι και πολυάριθμες οι συναντήσεις των σχεδόν εισηγητών. Ευχαριστώ θερμά την εισηγήτρια για την προσπάθειά της. Ήθελε το λόγο. Παρακαλώ. Ναι, πράγματι. Ε, δύο προτάσεις πάρα πολύ γρήγορα. Η κυρία Μιχάηλοβα είπε ότι πραγματικά δεν ήταν απλή η γνωμοδότηση η σύνταξη της νομοδότησης μας δυσκόλεψε γιατί υπήρχαν και άλλες επικαλύψεις ε, με την Επιτροπή Προπολογισμών, Επιτροπή Ελεκτού Προπολογισμού. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους κοιόδες εισηγητές αλλά και τους συνεργάτες, τους πολιτικούς συμβούλους και ιδιαίτερα το, τη γραμματεία για την ε, εξαιρετική υποστήριξη. Ήταν ε, καταπληκτική συνεργασία μας. Και παρά ε, το ότι είχαμε ένα πάρα πολύ στενό χρονοδιάγραμμα που εξακολουθεί να είναι στενό. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό το ότι έχουμε αυτή την πρώτη νομοδότηση πάρα πολύ καλή συμβολή. Θα παρακαλέσω βέβαια τους συναδέλφους ε, να προσέξουν ε, τι θα γίνει και στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Δηλαδή τελικά να μην ψηφίσουμε διαφορετικά σε κάποια σημεία στην Επιτροπή Προπολογισμών σε σχέση με το τι θα ψηφίσουμε σήμερα εδώ θα πρέπει να παραμένουμε σε επαγρύπνηση παρακαλώ τους συναδέλφους ε, αλλά ξέροντας πώς καλά συνεργαστήκαμε για την γνωμοδότηση δεν έχω και πολύ μεγάλη ανησυχία. Ευχαριστώ πάλι όλες και όλους. Σας ευχαριστούμε κύριε Κρέλ. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Η κυρία Κρέλ υπέβαλε τέσσερις ε, ευρύτατες συμβαστικές τροπολογίες ε, για τέσσερις παραγράφους, ε, για τέσσερα τμήματα του κειμένου μετά από συνεννόηση με τους σκιώδεις ηγητές. Αυτό να ληφθεί υπόψη στη μεθοδολογία της ψηφοφορίας. Θα είναι περίπλοκη η ψηφοφορία, γι' αυτό θα προσπαθήσω να μην βιάζομαι για να αποφύγω τα λάθη, αλλά διορθώστε με παρακαλώ αν υποπέσω σφάλματα. Ψηφίζουμε καταρχήν την τροπολογία 83. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Οπότε πάμε στη συμβιβαστική τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 92 τώρα. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 115. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 116. Ή μάλλον 120, συγγνώμη, 120. Τροπολογία 120. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 121. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 122. Υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Τροπολογία 140. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 141. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 157. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 158. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 159. Ποιος είναι... Α, συγγνώμη, είναι παρόμοια με την 158. Την αφήνουμε. 160. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 184. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 185 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 188 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 191 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 192 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 193 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 197 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 198 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 201 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 210. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 221. Ποιος είναι υπέρ της 221. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 222. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 226. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 227 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 231. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 232. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 233 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 235 ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 236 ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 237 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 240. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 240. Παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τροπολογία 241. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 242. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 243. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 245. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 247 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 248 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 251 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 261. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 262 με προφορική προσθήκη. Είναι κανείς κατά τις προφορικές τροπολογίες. Όχι, οπότε ψηφίζουμε μαζί με την προφορική τροπολογία 262. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 268. Σωστά. Ναι, 268. Ποιος είναι 269 μαζί για την επαρομοιότυπες υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Τροπολογία 270. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 271 με προφορική τροπολογία. Κύριε Μπούτα, έχετε να προσθέσετε κάτι, όχι. Είναι κανείς κατά της προφορικής τροπολογίας, υποβολής προφορικής τροπολογίας. Όχι, οπότε ψηφίζουμε τη 271 με την προφορική τροπολογία μαζί. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 27 τώρα για τις αιτιολογικές σκέψεις. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 28. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 31. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 33. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 48. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 58. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 68 ποιος είναι υπέρ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 4 έχει αποσυρθεί Τροπολογία 69, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, ή μάλλον καταπίπτει. Έχει εγκριθεί η συμβαστική 4. Οπότε πάμε στην τροπολογία 77. 77, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Τροπολογία 78, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 79, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 81 έχει αποσυρθεί. 82 τώρα. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε στην τελική ψηφοφορία. ηλεκτρονικά θα γίνει. Άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται μεγάλη διαφορά. Συγχαρητήρια κυρία Κρέλ. Και ευχαριστώ θερμά για τη βοήθειά σας στην ψηφοφορία. Συνεχίζουμε τώρα με την επόμενη έκθεση. Είναι η έκθεση που αφορά την τεχνική βοήθεια μάλλον μελλοντικές προοπτικές τεχνικής βοήθειας για την πολιτική συνοχής. Θέλετε να πείτε κάτι συνάδελφε, όχι. Ξεκινάμε λοιπόν. Τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχέσε εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχέσε εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχέσε εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχέσε ηλεκτρονική επαλήθευση. Τροπολογία 5 κοτσολίνο ηλεκτρονική επαλήθευση ε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας και απερίφθη. Συνεχίζουμε. Τροπολογία υπαριθμών 6 υπέρ. Κατά αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονική επαλήθευση από της τροπολογίας 6. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. Δεν το είχα διακρίνει αυτό το αποτέλεσμα. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω πως απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 40 υπέρ κατά αποχές νομίζω πως εγκρίνεται.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 Τροπολογία 64 υπέρ κατά αποχές. Καλύτερα ε, να κάνουμε και μια επαλήθευση. Ηλεκτρονική λοιπόν ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία από τις τροπολογίες 64. Πέρας. Και εγκρίνεται η τροπολογία. Τροπολογία 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 87. 87 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 89 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 90 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 91 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 92 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 93 υπέρ κατά αποχέσε εγκρίνεται. Και τώρα θα κάνουμε την τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Τόμασίτσε. Σας ευχαριστώ. Α, θέλετε να πείτε κάτι. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ήθελα να μιλήσω. Είναι ε, πριν, γιατί έπρεπε να ψηφίσω στην άλλη Επιτροπή Αλληλείας. Θα πω δύο λόγια τώρα για να ευχαριστήσω τους κοιόδης ε, εισηγητές ε, για την καλή συνεργασία. Είναι σαφές ότι όταν κάτι είναι πολύ σημαντικό, όλοι δουλεύουμε με ένα κοινό στόχο και τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Πολύ καλά τα πήγαμε και γρήγορα γρήγορα ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες και επομένως μπορούμε τώρα να συνεχίσουμε με την ημερήσια διάταξή μας ε, ε, η οποία προβλέπει ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά την έκθεση πρωτοβουλίας που αφορά την ανάπτυξη των μηχανισμών της πολιτικής συνοχής αναπεριφέρεια, ώστε να αντιμετωπιστούν οι δημογραφικές αλλαγές. Η συγγήτρια είναι η κυρία Γκαρθία Πέρες, Σήμερα θα μας δώσει μία γενική ε, ιδέα των ε, απόψεών της ε, και ενδεχομένως μετά θα ψηφίσουμε τον μήνα Σεπτέμβριο. Θα δώσω τον λόγο στην κυρία Πέρες και μετά στους Κιώδες. Κυρία Πέρες, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, λέει η κυρία Πέρες. Σήμερα Έχουμε την πρώτη συζήτηση, την πρώτη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας ε, που αφορά τις προκλήσεις ε, ε, των δημογραφικών αλλαγών που νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο και θα αποτελέσει κομβικό θέμα στις μελλοντικές μας συζητήσεις. Οι δημογραφικές αλλαγές είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τις πρόσφατες στατιστικές της της ε, Στατιστικής Υπηρεσίας ε, της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής δείχνει ότι γερνάει η Ευρώπη και κατά 19% θα αυξηθούν οι ηλικιωμένοι τα επόμενα χρόνια. Είναι επίσης σαφές ότι μέχρι το 2050 θα, θα επιβραδυνθεί ο βαθμός ανάπτυξης και θα, η επιβράδυνση αυτή θα είναι μεγαλύτερη από το 50 μέχρι το 70. Υπάρχουν πολλές περιοχές οι οποίες, στις οποίες ο πληθυσμός και γυράσκει ε, και μερικές φορές ε, σε ορισμένες περιπτώσεις ε, ο πληθυσμός μειώνεται. Υπάρχουν χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία και άλλες χώρες στις οποίες στις μητροπολιτικές περιοχές αυξάνει ο πληθυσμός ενώ στην Ήπεθρο μειώνεται. Και στην Ισπανία η κατάσταση είναι προβληματική. Σύμφωνα με τις τελευταίες τελευταίες στατιστικές ε, ε, πληροφορίες ε, το 50% των χωριών της Ισπανίας αντιμετωπίζουν κίνδυνο εξάλληψης. Στην Καστίγια Λεόν συζήτησα πάρα πολύ με τους υπεύθυνου το θέμα των δημογραφικών αλλαγών. Βλέπουμε ότι είναι πάρα πολλές οι περιφέρειες οι οποίες έχουν όλο και πιο ηλικιωμένους κατοίκους ε, όπου οι υπηρεσίες δεν υπάρχουν, ε, δεν υπάρχουν τράπεζες, δεν υπάρχουν σχολεία, δεν υπάρχει η δυνατότητα ιατρικής ε, φροντίδα, δεν υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει κανείς ασύρματες υπηρεσίες, ασύρματους τρόπους πληρωμής ή οποιαδήποτε άλλη δυνατότητα και πρέπει κανείς να πάει σε αυτές τις περιοχές για να δώσει χρήματα στους ανθρώπους ε, μιλάμε για περιοχές, ε, μιλάμε για ανθρώπους ε, που ζουν μονάχα απομονωμένοι και ακούνε μόνο τα, τα πουλιά και τα σπουργίτια και τίποτε άλλο, δεν έχουν καμία επαφή με τον έξω κόσμο και επομένως δεν έχουν καμία δυνατότητα να προσαρμοστούν στην συμπερίληψη την κοινωνική ή σε όποιες πρόοδους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν Υπάρχουν πάρα πολλά εδάφη και περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα απομονωτισμού κλπ. Ε, και αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Ε, θα πρέπει να ξαναβρεθεί αυτή η χαμένη και ιδιαίτερα περίπλοκη ισορροπία ανάμεσα στη, δημογραφία, στη δημογραφική εξέλιξη και στις περιφέρειες. Θα πρέπει να πούμε ότι η δημογραφική αλλαγή είναι ένα πρόβλημα ιδιαίτερο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντοπίζεται δε σε διάφορα στοιχεία. Ε, πρώτον, στην έλλειψη πυκνότητας. Ε, θα πρέπει λοιπόν ε, να βρεθεί μια λύση για αυτές τις περιφέρειες με ιδιαίτερα χαμηλή πυκνότητα. Και επίσης έχουμε περιφέρειες οι οποίες πάντα είχαν χαμηλότερη πυκνότητα, αλλά και περιφέρειες στις οποίες διαρκώς μειώνεται η πυκνότητα αυτή. Δεύτερη πρόκληση, ε, πολύ σημαντική επίσης, είναι η γύρανση του πληθυσμού. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, πρόκειται για γνωστό δημογραφικό ε, ε, γεγονός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως, εν μέρη, πρόκειται για μια φυσιολογική δημογραφική αλλαγή, αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι έχει ενταθεί το πρόβλημα αυτό. Τρίτο πρόβλημα είναι η μείωση της γεννητικότητας. Έχουμε λιγότερους νέους και λιγότερα ε, μικρά παιδιά. Θα πρέπει μέσω πρόθεσμα οπωσδήποτε να αλλάξουν και οι σχέσεις όσον αφορά την οικογένεια και τη δυνατότητα παροχής βοήθειας στις ε, οικογένειες με μικρά παιδιά. Ε, το ε, επόμενο ε, θέμα είναι η απομάκρυνση και ο απομονωτισμός που στην ουσία είναι αποτέλεσμα όλων των προηγουμένων στοιχείων. Βεβαίως και λόγω των μεταναστευτικών μετακινήσεων σε μερισμένες περιπτώσεις οι δημογραφικές αλλαγές γίνονται πιο έντονες. Οι δημογραφικές αλλαγές υπήρχαν πάντα αλλά η έντασή τους είναι πρωτοφανής. Υπάρχουν Υπάρχουν περιοχές επίσης στις οποίες, ε, ε, ε, στις οποίες συνυπάρχουν όλες οι αναφορές, που, όλοι, όλοι οι λόγοι που ανέφερα προηγουμένως. Επίσης σε όλες τις προηγούμενες αιτίες που ανέφερα, σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να προσθεθεί και το θέμα της διαφοροποίησης, της ανισορροπίας των φύλων. Γιατί στην περίπτωση των χωριών που ανέφερα προηγουμένως υπάρχει και έλλειψη γυναικείου πληθυσμού που είναι η βάση για να αναπτυχθεί ο πληθυσμός. Μέχρι τώρα πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει γενική ευρωπαϊκή στρατηγική για να εντοπιστεί αυτή η πρόκληση. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει υπόψη ε, το δημογραφικό στοιχείο σε όλες τις στρατηγικές και όλες τις πολιτικές, ε, στους προϋπολογισμούς ε, και σε όλους τους προσανατολισμούς που αφορούν ανάπτυξη νέων πολιτικών, κυρίως όσον αφορά περιβαλλοντικές, εργασιακές, αγροτικές πολιτικές. Θα πρέπει να ε, σκύψει πάνω στο θέμα της δημοκρατικής αλλαγής ε, έτσι όπως, η Ευρωπαϊκή, έτσι όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη ζήτησε από το Σεπτέμβριο του 2015. Θέλουμε ε, επίσης αξιοπρεπή εργασία, καλές συνθήκες εργασίας, περιφερειακές στρατηγικές προώθησης της απασχόλησης. Η αλλαγή μοντέλου και υποδείγματος θα πρέπει να ληφθεί υπόψη έτσι ώστε ώστε να αλλάξει η όψη των περιφερειών. Θα πρέπει να υπάρχουν ανταγωνιστικές τιμές ε, σε περιφέρειες με λιγότερη πυκνότητα πληθυσμού οι δημόσιες ε, υπηρεσίες, ε, οι τοπικές, ε, οι τοπικές, τα τοπικά μέσα επικοινωνίας και μεταφοράς, η δυνατότητα να ενταχθούν μετανάστες, επίσης και κάποια νέα στοιχεία που θα κάνουν πιο ελκυστική την Ήπεθρο, θα πρέπει να αποτελέσουν κεντρικά θέματα της αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα σοβαρά και ε, διαρκή προβλήματα της ε, δημογραφικής ε, αλλαγής. Ανέφερα προηγουμένως τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πυρωτικές ζώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, βλέπουμε ότι και σε άλλες περιφέρειες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα και συγκριτικά μειονεκτήματα πρέπει οπωσδήποτε να βοηθηθούν. Επίσης θα πρέπει να βρεθούν νέα κριτήρια ε, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα ε, προβλήματα, τα δημογραφικά, τα οποία αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα, ε, ιδιαίτερες περιοχές. Όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν περιοχές οι οποίες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα και όσον αφορά την πυκνότητα του πληθυσμού και όσον αφορά το ΑΕΠ, αυτές οι περιοχές κατά προτεραιότητα θα πρέπει να βοηθηθούν ε, με ευρωπαϊκά ε, κονδύλια. Ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν αρκετά κονδύλια έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι δημογραφικές αλλαγές. Τα διορθωτικά ταμεία, τα κοινωνικά ταμεία θα πρέπει ιδιαίτερως να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις των δημογραφικών αλλαγών. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τις περιοχές που έχουν σημαντικά δημογραφικά μειονεκτήματα και ε, να ληφθούν ιδιαίτερε υπόψη ανάγκε του στα υπάρχοντα ταμεία. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το 2020 θα πρέπει να περιλαμβάνει και μια εμβληματική πρωτοβουλία για τα δημογραφικά ζητήματα. Και μάλιστα οι περιοχέ με δημογραφικέ ε, προκλήσει, που αντιμετωπίζουν δημογραφικέ προκλήσει, θα μπορούσαν να επωφεληθούν από μια τέτοια πρωτοβουλία που θα μπορούσαμε να την αποκαλέσουμε πληθυσμό ε, και κυρίω να επικεντρωθούμε σε τρει κατηγορίες στην ανάπτυξη που θα είναι ευφυής, ε, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς. Και μάλιστα το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020 θα πρέπει να δώσει μια όθηση ώστε να αντιμετωπιστούν οι δημογραφικές προκλήσεις και φυσικά είναι απαραίτητο κάτι που ήδη έχουμε διεκδικήσει πολλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον καλύτερο συντονισμό και την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων εργαλείων και μηχανισμών που διαθέτουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την κοινή γεωργική πολιτική, τα διαρθρωτικά ταμεία και τα ευρωπαϊκά επενδυτικά ταμεία, ώστε να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπό του ε, στι δημογραφικέ αλλαγέ. Όλα αυτά είναι ζητήματα που αποτέλεσαν τη βάση για την έναρξη της ε, εργασιών εκπόνησης αυτής της πρωτοβουλίας, ε, της έκθεσης πρωτοβουλίας αλλά φυσικά περιμένω και τις απόψεις των συναδέλφων, περιμένω τις ε, προτάσεις σας για θέματα που θέλετε να συμπεριλάβουμε στην έκθεση πρωτοβουλίας και ευελπιστώ ότι και στις μελλοντικέ μας συναντήσεις και συζητήσεις ε, θα καταφέρουμε να διαμορφώσουμε μια έκθεση που θα μας δώσει όθηση προκειμένου να αντιμετωπίσουμε και τις μελλοντικές συζητήσεις για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και περιμένω και εγώ ανυπόμονα τις δικές σας προτάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για τις αρχικές σας σκέψεις και τώρα θα συνεχίσουμε με ε, τις παρεμβάσεις εκ μέρους ε, των σχεδόν. Ο κύριος ε, Βαλκάρθελ έχει πρώτα απ' όλα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πράγματι, η Ευρώπη σήμερα αντιμετωπίζει αυτό το σοκ ε, της διαφορικής δημογραφικής ανάπτυξης. Ε, δηλαδή, ενώ αυξάνεται στον υπόλοιπο κόσμο πληθυσμός και υπάρχουν όλο και περισσότεροι νέοι, ε, στην περίπτωση της Ευρώπης ο πληθυσμός και μειώνεται και γυράσκει. Και αυτό σίγουρα δίνει το νόημα και το περιεχόμενο σε αυτήν την έκθεση. Πρέπει δηλαδή να προωθήσουμε μακροπρόθεσμα προγράμματα και σχέδια έξω και επικροτώ ιδιαίτερα την πρόοδο που συνιστά η έκθεση αυτή. Η δημογραφική πρόκληση είναι πάρα πολύ οξυμένη και ιδίω όπως υπόθηκε σε περιφέρειες της Ισπανίας, όπως είναι η Καστιλεόν για παράδειγμα, η Γαλλικία, Αστούρια, Καστίγια Λαμάντσα, η, η Αραγωνία και θα πρέπει να δώσουμε μια απάντηση όχι μόνο για αυτές τις περιφέρειες, αλλά για όλους. Ή όλες τις περιφέρειες μπορεί να μένει πίσω ε, μια περιοχή, μια περιφέρεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι χάνει μόνο αυτή η περιοχή, αυτή η περιφέρεια, αλλά ολόκληρη Ευρώπη. Γι' αυτό πρέπει να σημειώσουμε κάποια πρόοδο. Ό,τι αφορά τώρα τη μεταρρύθμιση τη πολιτική συνοχή, οι δημογραφικέ προκλήσει θα πρέπει να ληφθούν πολύ περισσότερο υπόψη, κατά την άποψή μα. Το 2016 ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έναν οδικό χάρτη που θα μα επέτρεπε να προχωρήσουμε πιο πέρα. Να μην έχουμε μόνο δείκτη το ΑΕΠ. Θέλαμε ε, να έχουμε και ε, άλλου δείκτε για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις, όπως είναι η διασπορά του πληθυσμού μεταξύ αυτών των αναπτυξιακών δικτών. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι περιοχέ που αντιμετωπίζουν δημογραφικέ απορρίψει συνήθω αναπτύσσονται λιγότερο από το μέσο όρο και όπω είπε και η συγγήτρια, αντιμετωπίζουν περισσότερε δυσκολίε σε ό,τι αφορά την παροχή υπηρεσιών στου πολίτε. Θα πρότεινα ορισμένες ε, Σκέψεις πρώτα απ' όλα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη διασυνδέσεων ε, για απόμακρες ή αεροκατοικημένες περιοχές με βελτίωση της πρόσβασης στο διαδίκτυο. Δεν χωρεί αμφιβολία ότι η, διασύνδεση, η συνδεσιμότητα της υπαίθρου είναι κάτι πολύ σημαντικό για τους νέους επαγγελματίες για να μπορούν να, να αναπτύσσουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, επιχειρηματικές δραστηριότητες στην υπαίθρο. Πολύ σημαντικό είναι ο ρόλος της υπαίθρου επίσης σε τομείς όπως είναι ο οικολογικός τουρισμός ή το ηλεκτρονικό εμπόριο. Για αν εκμεταλλευτούμε αυτού του κλάδου, θα πρέπει να προωθήσουμε την καινοτομία που θα τονάσει περισσότερο τι τοπικέ οικονομίε και θα αναζωογονήσει παραδοσιακά επαγγέλματα και επιτιδεύματα. Θα πρότεινα ε, η συγκεκριά να συμπεριλάβει αυτά που είπα, διότι δεν είναι σημαντική μόνο η δημογραφική ανάπτυξη, αλλά ε, στο χρόνο, αλλά και στο χώρο, γιατί οι νέοι φεύγουν και παραμένουν οι πιο ηλικιωμένοι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ε, στις πόλεις να αυξάνεται σημαντικά ε, η ε, τιμή, να αυξάνονται οι τιμές και το βετικό επίπεδο πιο ακριβό, το αντίθετο να γίνεται στην Ήπεθρο. Είναι σημαντικό λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τις δημογραφικές προκλήσεις αν θέλουμε να διατηρήσουμε και το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο το οποίο εδράζεται στην αλληλεγγύη τη δεγενειακή, αλλά και στην αλληλεγγύη μεταξύ εδαφών, μεταξύ περιφερειών. Ακριβώ σε ό,τι αφορά τη δεγενειακή αλληλεγγύη. Αυτό θα πρέπει να παραμείνει παρά τι δημογραφικέ ανισορροπίε. Θα πρέπει να ζητήσουμε νέε χρηματοοικονομικέ ισορροπίε. Και η δαφική ισορροπία θα πρέπει στόχο ε, να έχει να κλείσει το χάσμα μεταξύ αυτών των περιοχών που παράγουν πλούτο και αυτών που χρησιμοποιούν τι κοινωνικέ υπηρεσίε. Επομένω, θα πρέπει να δοθεί μια ευρεία συντονισμένη απάντηση, όπω ζητά και η Επιτροπή των Περιφερειών στην γνωμοδότηση χρηματοδότησή της για τις δημογραφικές προκλήσεις. Ε, κυρία Πρόεδρε, ήταν ε, σκόπιμο να το πούμε, ε, δεν υπάρχει κανένας καλύτερος από τους περιφερειακούς διαχειριστές. Θα μας πει πώς είναι η κατάσταση επιτόπου. Θα πρέπει να τονίσουμε και την ευφύ εξειδίκευση πρέπει να στοιχηματίσουμε υπέρ της καινοτομίας, της έρευνας. Οι στρατικές αυτές θα δώσουν στις περιφέρειες τη δυνατότητα να γίνουν ανταγωνιστικοί πόλη, ανταγωνιστικό. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να εξηγήσουμε στους πολίτες μας ότι μια ένωση που μπορεί να παράγει ανάπτυξη και απασχόληση είναι αναμφίβολα το καλύτερο περιβάλλον, το καλύτερο πλαίσιο για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων και μεταξύ αυτών τη δημογραφική πρόκληση. Αυτή η έκθεση μπορεί να το καταδείξει υποστηρίζοντα ένα πραγματικό κοινωνικό θεματολόγιο που θα αναφέρονται σαφώ οι δημογραφικέ προκλήσει και θα υποστηρίζεται ένα αναπτυξιακό μοντέλο που δεν θα αφήσει κανέναν πίσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρος. Πορέμπα, δεν είναι εδώ. Γιάκοφτσιτς, επόμενος κοιόδης, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να κάνω και εγώ κάποια σύντομα σχόλια. Έχοντας υπόψη ότι το θέμα αυτό ε, ιδιαίτερα τα τελευταία 25 χρόνια που ασχολούμαι με αυτή την πολιτική, το ζήτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ήταν ανέκαθε σημαντικό για την Κροατία και πριν την ε, προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ θα ήθελα να σταθώ σε δύο κυρίως σημεία, σε δύο θέματα που τόνισε και η συγγήτρια. Ε, το βασικό θέμα είναι η γύραση του πληθυσμού. Και φαίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα έχουμε μια Ήπειρο που θα αποτελείται κυρίως από ηλικιωμένους στο μέλλον. Και ε, σε πολλές χώρες θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα πώς θα πληρώνουν τις συντάξεις, γιατί θα είναι μεγαλύτερο το ποσοστό των ηλικιωμένων. Αυτό το θέμα λοιπόν της γύρεσης του πληθυσμού είναι πολύ σημαντικό και σίγουρα το φαινόμενο θα οξυθεί στο μέλλον. Οπότε αυτό το θέμα θα πρέπει να μας απασχολήσει και να δούμε κατά πόσο έχουμε τη δυνατότητα να βρούμε κάποιες κοινέ λύσεις, κάποιους κοινούς τρόπους ε, ε, να αντιμετωπίσουμε το θέμα της γύρανσης του πληθυσμού, δεδομένης της διαφοράς των συνταξιοδοτικών μας συστημάτων. Πάντως το θέμα της γύρανσης του πληθυσμού θα πειράσει όλες τις χώρες και θα μας απασχολεί όλο και περισσότερο στο μέλλον. Και επειδή υπάρχει αλληλεξάρτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα αυξηθεί παντού αυτό το ζήτημα. Επίσης, ε, ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τα ζητήματα της ανάπτυξης πέθρου και ξέρω ότι στην Κροατία είναι πολύ σημαντική αυτή η πρόκληση, αλλά υπάρχουν λύσεις. Και δεν θα ήθελα να επαναλάβω αυτά που είπε η συγγήτρια, γιατί πραγματικά κατέθεσε προτάσεις ε, πολύ εύστοχες. Τώρα, δεν είμαι σίγουρος αν χρειαζόμαστε ιδιαίτερο ταμείο για κάτι τέτοιο, αυτό θα το συζητήσουμε, γιατί έχουμε πολλά ταμεία. Το βασικό όμω είναι το περιεχόμενο, η ουσία. Δεν είναι το θέμα του τύπου αν θα έχουμε ξεχωριστό ταμείο ή όχι. Το θέμα είναι πώς θα βρούμε αυτά τα χρήματα και πώς θα τα επενδύσουμε σωστά στην Ήπεθρο. Γιατί η Ήπεθρος ιδιαίτερα στην Μεσόγειο, γιατί ακούσαμε τα προβλήματα στην Ισπανία, αλλά και στην Κροατία έχουμε παρόμοια προβλήματα και στην Ιταλία έχουμε ε, παρόμοια προβλήματα. Οπότε ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσογείου η Ήπεθρος ε, αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα, γι' αυτό και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και φροντίδας, πολύ περισσότερο από ό,τι σήμερα. Και αυτή την άποψη είναι πολύ σωστά διαρθρωμένη αυτή η έκθεση με βάση αυτά που μας είπε η εισηγήτρια και πιστεύω ότι θα πρέπει να βρούμε κάποιες απαντήσεις στα καυτά αυτά ερωτήματα γιατί υπάρχουν πολλοί αρνητικές δημογραφικές διαδικασίες και εξελίξεις που θα συνεχιστούν δυστυχώς δεν πρέπει να έχουμε ψευδεστήσεις, θα συνεχιστεί αυτή η αρνητική δημογραφική εξέλιξη, θα πρέπει λοιπόν να βρούμε κάποιες λύσεις και νομίζω ότι έτσι θα καταφέρουμε να σημειώσουμε ένα βήμα πρόοδου. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Δεν βλέπω την κυρία Βαλίνα. Υπάρχει κάποιο άλλο που θα ήθελε το λόγο εκ μέρου τη κυρία Βαλίνα πρώτα, Βαλίνα πρώτα απ' όλα, όχι. Ρόπε ή εκ μέρου τη Ρόπε, κυρία Βάνα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Μιλώ εδώ εξ ονόματος του κύριου Ρόπε που έστειλε κάποιες σημειώσεις τις οποίες και θα αναγνώσω μεταξύ των προκλήσεων που αντιμετωπίζει επί του Ευρωπαϊκή Ένωση το δημογραφικό στοιχείο ίσως είναι το πιο αποτιμημένο η σημαντική ε, αύξηση ε, του πληθυσμού σε 1.300 δήμους και πάνω από 11.000 κοινότητες βλέπουμε ότι δεν είναι πραγματικότητα, μειώνεται ο πληθυσμός και γυράσκει. Αυτό σημαίνει και με λιγότερη όθηση στην οικονομική ανάπτυξη και λιγότερη έμφαση στην κοινωνική πρόνοια. Θα πρέπει να επιτύχουμε τους στόχους της εδαφικής κοινωνικής συνοχής, άρα να βελτιώσουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο, να έχουμε καλύτερες ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών και να προσανατολίσουμε έτσι τα δευτικά τα οι θέσεις εργασίας να είναι και εκτός ε, ε, πόλεων και να έχουμε καλύτερες θέσεις εργασίας για νέους ηλικιωμένους γυναίκες. Επίσης, θα πρέπει να αλλάξουμε αιστεία στην πολιτική συνοχή, να μην έχουμε μία ε, προσέγγιση που θα έχει να κάνει μόνο με το πώ εφαρμό, που πηγαίνουν αυτά τα κονδύλια, αλλά θα πρέπει να δούμε τη βιωσιμότητα, η μακροβιότητα τη απασχόληση και τη κοινωνική συνοχή. Είμαστε υπέρ τη εξέβρισης σωστή ισορροπία μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών και προσβλέπω στη συνεργασία με την εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε Ανταμάτο. Grazie. Είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει ιδιαίτερος πρέπει να σας ομολογήσω. Και ε, περιμένοντας το προσχέδιο της έκθεσης ε, μπορώ να κάνω κάποιες γενικές σκέψεις. Ε, ε, είναι πολλές ε, οι ε, μελέτες οι οποίες υπογραμμίζουν ε, την διαρκώς και μεγαλύτερη τάση μείωσης του πληθυσμού και βεβαίως αυτό επιδεινώνεται σε συγκεκριμένες περιφέρειες, ας πούμε σε ορισμένες περιφέρειες οι οποίες είναι οι διαγραφομακρυσμένες, οι ορεινές, της υπαίθρου, οι ιδιαίτερα περιφερειακές κλπ. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ε, αυτό το δημογραφικό πρόβλημα το οποίο μαζί με τα οικονομικά προβλήματα και τα κοινωνικά προβλήματα ε, μπορούν να οδηγήσουν συγκεκριμένες περιφέρειες σε μεγάλη φύση, σε μεγάλη ε, μείωση του πληθυσμού τους και σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Θα πρέπει οπωσδήποτε οι πολιτικές οι οποίες αφορούν την οικογένεια, την εκπαίδευση, την παροχή ιατρικής φροντίδας να ληφθούν υπόψη. Γι' αυτό λοιπόν ε, νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία της έκθεσης Σιώτοβα ε, για τις ορεινές περιοχές. Εκεί ζητούσαμε ε, επιπλέον κίνητρα έτσι ώστε μικρές μεταποιητικές βιομηχανίες και μικρές αγροτικές επιχειρήσεις στις ορεινές περιοχές να βοηθηθούν με συγκεκριμένα επιπλέον κίνητρα. Γιατί εάν θέλουμε να διατηρήσουμε ένα ίδιο επίπεδο ποιοτικό, οπωσδήποτε ε, ε, θα πρέπει οι προσπάθειες που θα καταβληθούν σε αυτές τις ε, επιχειρήσεις και σε αυτές τις περιοχές να είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι σε άλλες παιδινές περιοχές. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη και οι βιοτεχνικές δραστηριότητες σε απομακρυσμένα χωριά και ορεινά χωριά με φθήνοντα πληθυσμό. Ε, επίσης ε, προέκυψε πάλι ε, στην Ιταλία το πρόβλημα αυτό όπου κατεδείχθη ότι όχι μονάχα σε απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές, αλλά και σε πιο παιδινές ε, έχουμε μεγάλη μείωση του πληθυσμού, πράγμα που σημαίνει ότι ε, ε, οι δραστηριότητες, οι αγροτικές εγκαταλείπτονται, εγκαταλείπονται και επίσης είναι, χώρες, είναι περιφέρειες οι οποίες πρέπει να βοηθηθούν οπωσδήποτε. Αυτός είναι, αυτό είναι ένα είδος σεισμού, ένας άλλος σεισμός είναι ε, αυτός που συνέβη στην ε, Αματρίτσα ας πούμε. Ε, πρόκειται για περιφέρειες οι οποίες έχουν καταστραφεί εντελώς και οι οποίες θα πρέπει οπωσδήποτε να βοηθηθούν. Εμείς σαν κίνημα των πέντε αστέρων θα βοηθήσουμε αυτές τις περιοχές γιατί θα πρέπει οπωσδήποτε να βοηθηθούν και θα πρέπει οπωσδήποτε να υπογραμμιστεί το πρόβλημά τους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Έχω εδώ ένα κατάλογο με 7 αγορητές. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Βέστηφαν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όλα όσα ανέφερε μόλις πριν η συγγήτρια μπορώ να τα υπογραμμίσω και εγώ και να συμφωνήσω Είχαμε και την έκθεση του 2011 για τη αλλαγή και τι ε, μέσα ε, θα χρειαστούν για την αντιμετώπιση αυτών των ε, αλλαγών. Η δημογραφία και αυτή η αλλαγή δημογραφική μπορεί να αποτελέσει και ευκαιρία. Απλά θα πρέπει να υπάρξει χρηματοδότηση, θα πρέπει να την καθοδηγήσουμε σωστά, το είπε και η συγγήτρια. Θα ήθελα να αναφερθώ λοιπόν και στη δική μου έκθεση και για τα βασικά ε, συστατικά στοιχεία της πολιτικής συνοχής. Αναφέρω λοιπόν συγκεκριμένα ότι σε ό,τι αφορά τη μέθοδο ε, και την ε, κατάσταση της ανάπτυξης, αυτό στο μέλλον θα παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο μέλλον για τις περιφέρειες και επίσης η η ευελιξία, ελαστικοποίηση τη χρηματοδότηση είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προωθήσουμε. Όμω θα ήθελα να ε, προειδοποιήσω. Μιλήσαμε και μιλούμε πολύ για την υπεθρο για τι αγροτικέ περιοχέ. Γνωρίζω πολύ καλά ότι σε ό,τι αφορά τη δημογραφία πράγματι φεύγουν από την Ήπεθρο οι νέοι. Γι' αυτό και είχαμε πει και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο θα πρέπει να ε, υιοθετήσουμε κάποιες νέε δόμε. Γιατί δική μου την περιφέρεια μπορώ να πω και ξέρω ότι ισχύει και για άλλε περιφέρειε περιφέρειες ότι υπάρχουν επιχειρησιακά προγράμματα που έχουν δρομολογηθεί. Αυτό δεν είναι παρά μια αρχή. Είναι όμως κάτι που πρέπει να γίνει, θα πρέπει να ενισχυθεί. Προειδοποιώ όμως ε, και σε σχέση με αυτή τη συζήτηση θα πρέπει ε, να μην κάνουμε μία διάκριση μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών, να μην τις φέρουμε σε αντιπαράθεση. Δηλαδή υπάρχουν διαφορές, αλλά θα πρέπει να συνεργαστούμε και να αντιμετωπίσουμε από κοινού τα προβλήματα τα δημογραφικά και τις ανισότητες που προκύπτουν θα πρέπει να τις εξαλείψουμε κατά το δυνατόν. Ε, η έκθεση αναφέρει πολύ καλά σημεία. Είναι πάρα πολύ καλό να ε, πιστεύω να έχουμε αναφορές σχετικά με αυτά τα θέματα και να καταδείξουμε πόσο σημαντικό είναι για μας, για τους πολίτες ε, και πραγματικά και στην Ήπεθρο να μπορεί να ζει ο κόσμος καλά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Βανίλ Στερόι. <clears throat> Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι εξαιρετική η πρόταση της συγγήτριας ε, για ανάλυση αυτού του θέματος. Είδαμε τις ραγδαίες εξελίξεις στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχαμε ένα αποκαδεκατισμό του πληθυσμού και τώρα θα πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό. Ε, σε τι κατάσταση βρίσκεται ο πληθυσμός μας, τι γίνεται με τη γενετικότητα, γεννιούνται παιδιά, γιατί θα πρέπει να φτάσουμε στα 2,2 παιδιά ένα ζευγάρι για να επιβιώσουμε, για να διατηρήσουμε δηλαδή ε, μια βιώσιμη δυναμική και ένα κατάλληλο το πληθυσμού. Στην Ιταλία βρισκόμαστε στο 1,6 ακόμη και υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σίγουρα οι αλλαγές θα ενισχυθούν και οι διαφορές ε, θα μεγαλώσουν δεν μπορεί να μας αφήνει διάφορους αυτό το θέμα. Θα πρέπει να το αναλύσουμε ενδελεχώς και να αναζητήσουμε και λύσεις. Επίσης, έχουμε παιδινές περιοχές ή ε, αγροτικές ζώνες, ε, ε, την Ήπεθρο, με ιδιαίτερες ανάγκες. Μέχρι στιγμής τα μέτρα μας ήταν αντιπαραγωγικά, γιατί εθαρρύναμε τους νέους να εγκαταλείψουν την Ήπεθρο και ενισχύσαμε αυτή την αστιφιλία. Τώρα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες των μέτρων που υιοθετήσαμε. Αντί να έχουμε μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων, θα πρέπει να επινοήσουμε μια Ευρώπη που να επιτρέπει σε όλους να προοδεύουν ταυτόχρονα και να μην ε, προσελκύονται οι νέοι από τις πιο ε, ευημερούς περιοχές, ε, να μην έχουν κίνητρα να εγκαταλείπουν τα χωριά και τις πόλεις τους Αναζητώντα ένα καλύτερο μέλλον. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ευνοϊκέ συνθήκες παντού. Επίσης έχουμε νέα ταμεία, νέους μηχανισμούς. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα ε, τα συνδυάσουμε με τα υφιστάμενα ταμεία και τους υπάρχοντες μηχανισμούς. Να επενδύσουμε επίσης στην παιδεία, στη δημιουργία θέσεων απασχόληση, στην επικοινωνία, την ψηφιοποίηση, τη διασυνδεσιμότητα, πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη, πρόσβαση ακόμη και στην ηλεκτρονική υγεία. Θα πρέπει να βρούμε συνολικές λύσεις. Το είπαμε και στην προηγούμενη έκθεση για τα δομικά στοιχεία της συνοχής μετά το 2020. Επίσης αναφερθήκαμε και στο άρθρο 63. και κάναμε έναν απολογισμό της κατάστασης σε εθνικό επίπεδο. Είχαμε ήδη πει λοιπόν από τότε ότι οι δημογραφικές αλλαγές θα πρέπει να είναι από τα κριτήρια που θα λαμβάνουμε υπόψη κατά την εφαρμογή των ε, ταμείων. Το ΑΕΠ είναι χρήσιμο κριτήριο, αλλά θα πρέπει να είναι το μοναδικό, γιατί τα τελευταία χρόνια είχαμε μείωση του ΑΕΠ και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι θα αλλάξει η κατάσταση. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε μέτρα και να δημιουργήσουμε νέες προοπτικές για να επιτρέψουμε στον κόσμο να παραμείνει στην Ήπεθρο. Και σίγουρα θα πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό και να καταμετρήσουμε τις ε, συνέπειες των ε, μέτρων μας. Και ήταν εξαιρετική και η έκθεση Westphal, γιατί μας ε, επέτρεψε να καταλήξουμε σε ένα πλαίσιο συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλους τους ενδιαφερόμενους πολιτικής αυτής. Μιλήσαμε επίσης για την ενεργό είχαμε επαφή με εκπροσώπους της βιομηχανίας, του τομέα της υγείας, τοπικούς και περιφερειακούς ε, φορείς. Θα πρέπει να εμπλέξουμε όλους αυτούς τους ενδιαφερόμενους και να καταλήξουμε σε συνέργειες. Επίσης μιλήσατε για την εκδήλωση της 29ης Απριλίου που είναι η μέρα της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών. Επίσης, πέμπτη το πρωί θα έχουμε και πρόγευμα εργασίας με θέμα την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Οπότε θα ήθελα να καλέσω και την ε, εισηγητριακή για να παρακολουθήσει την παρουσίαση των σχεδίων που θα υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που είναι ε, παραδείγματα προς ε, από διάφορες ευρωπαϊκές περιφέρειες. Θα πρέπει επίσης να δημιουργήσουμε θετικές ευκαιρίες και προοπτικές οικονομικές, όχι μόνο για τους νέους, αλλά και για τους ηλικιωμένους, για τους πρεσβύτερους. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε τα τοπικά και περιφερειακά προβλήματα, όπως ε, την ανεργία που είναι από τις βασικές μάστιγες. Είχαμε μια νέα πρωτοβουλία με ένα πιλωτικό πρόγραμμα στην Επιτροπή Γεωργίας για την έξυπνη ανάπτυξη στην Ήπεθρο και μάλιστα οι Επίτροποι Χόγκαν και Κρέτσου παρουσίασαν αυτό το σχέδιο των ε, έξυπνων κοινοτήτων. Αυτό είναι ένα παράδειγμα του δυναμικού που έχουμε και της, ε, των επιτεγμάτων που μπορούμε να επιτύχουμε σε θέματα απασχόλησης και παροχής υπηρεσιών. Το σχέδιο αυτό λοιπόν είναι αξιέπαινο και θεωρώ ότι είναι πολύ εύστοχα το σχόλιο που μας έκανε η εισηγήτρια. Θα πρέπει να βρούμε απτές λύσεις για να κινητοποιήσουμε τα περιφερειακά διαρθρωτικά και επενδυτικά μας ταμεία. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μπόκοβιτς, ευχαριστώ πολύ. Πολύ σημαντικό το θέμα ε, και χαίρομαι που περιλαμβάνει η έκθεση πολλά σημαντικά ζητήματα. Πράγματι γυράζει και ο πληθυσμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδίω στην Ευρώπη, ε, μιλώντας στην Ήπεθρο. Και Αναφέρθηκε επίσης ότι εγκαταλείπουν την Ήπεθρο οι νέοι και μετακινούνται στις πόλεις, σε αστικές περιοχές. Αυτό δίνει έμφαση επίσης και στη μετανάστευση, ε, στην έκθεση μάλλον δίνεται έμφαση και στη μετανάστευση μεταξύ, στις μετακινήσεις ε, μεταξύ των κρατών μελών. όπου Υπάρχει πληθυσμό που μετακινείται στι ε, χώρε με ταχύω αναπτυνόμενε οικονομίε. Ε, πρέπει να μετωπίσουμε τι προκλήσει ε, και την αλλαγή τη σύνθεση του πληθυσμού. Δεν έχει ανταποκριθεί μέχρι στιγμή με σωστού ρυθμού η πολιτική συνοχή ούτε οι πολιτικέ. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε τι απαραίτητε υποδομέ για να εξασφαλίσουν ε, ένα αξιοπρεπέ βιωτικό επίπεδο στον 21ο αιώνα, τηλεπικοινωνίες, περιβάλλον, μεταφορέ, παιδεία, υποδομέ, κοινωνικέ μεταξύ άλλων υποδομές, υγεία, αθλητισμός κτλ. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Είμαι από τη Σλοβενία που είναι μία από τις χώρες που είχε ε, προωθήσει μια απο τι χώρε πολιτική ανάπτυξης. Αυτό ανάπτυξη. αυτο από τη δεκαετία του 70 που ήμασταν μια σοσιαλιστική χώρα. Δύο εκατομμύρια είναι οι κάτοικοι ο ε, πληθυσμό τη χώρα μα ε, και αυτή την πολυκεντρική προσέγγιση ε, την έχουμε για το Μάριμπορ, τη Λουμπλιάνα και άλλε πέντε μεγάλες περιφέρειες. Αφενό και άλλα 35 μικρότερα αναπτυξιακά κέντρα στη Σλοβενία. Με την πολιτική αυτή ο κόσμος παρέμεινε στην Ήπεθρο. Ζει και εργάζεται στην Ήπεθρο. Και νομίζω ότι θα πρέπει αυτή η πολιτική να βρει μιμητές και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, στη χώρα μου πάνω από το 50% του πληθυσμού εξαπλήθηκε να παραμείνει σε αγροτικέ περιοχέ. Είμαστε η μόνη χώρα. Έχουμε χρησιμοποιήσει και προ το σκοπό αυτό για την δημιουργία δηλαδή, των σχετικών υποδομών και τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να θέλουν οι νέοι να μείνουν στην υπαίθρα της αγροτικές περιοχέ, αλλά πρέπει να τους δώσουμε δουλειέ. Ε, και αυτή είναι μια σημαντική πρόκληση. Θέλω να υποστηρίξω αυτό που είπε ο κ. Βανίστελ Ρόι Πώς δηλαδή θα αξιοποιήσουμε το δυναμικό, ε, τις δυνατότητες της σημερινής γενιάς ε, να μην αντιμετωπίζονται ως βάρος και το ίδιο και με τους ηλικιωμένους πρέπει να συμβεί. Στη Λοβενία έχουμε ένα έργο, ένα πρόγραμμα όπου υπάρχουν ε, ηλικιωμένοι που βοηθούν άλλους ηλικιωμένους, πιο νέοι συνταξιούχοι, εντός αγωγικών βοηθούν πιο ηλικιωμένους συνταξιούχους ώστε να έχουμε ποιοτική ζωή. Υπάρχει λοιπόν αυτή η συνεργασία με των γενών, κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Και εγώ έχω ξεκινήσει ένα project και πριν από 40 ημέρες οργανώσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα πάρα πολύ καλό σεμινάριο παρουσία των επιτρόπων Γκρέτσου Χόγκαν ε, για τα μικρά χωριά. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μεγάλες προκλήσεις. Τεχνολογική επανάσταση που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Αυτό δεν θα πρέπει να αποβεί σε βάρος των μικρότερων χωριών. Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να αξιοποιηθούν με πάρα πολύ καλό τρόπο και στις αγροτικές περιοχές, όσο αφορά το εμπόριο, τον τουρισμό ή στον τομέα των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών. Θα προσπαθήσω δεν να καταρτήσω και ένα πιλωτικό πρόγραμμα σχετικά. Πρέπει να σκεφτούμε και το ενδεχόμενο να έχουμε τα εργομέφη χωριά ε, στις επόμενες προσωπικές προοπτικές, ώστε να παραμείνει υπεθρός, ελκυστικός τόπος πάνω για τους νέους και στο μέλλον. Ποιος έχει όμως την ευθύνη εδώ, αυτό είναι ένα σημαντικό ερώτημα. Η αρχή της επικουρικότητας νομίζω δεν είναι κάτι που θα πρέπει να σεβαστούμε. Πρώτα απ' όλα οι δήμοι, οι κοινότητες, μετά οι περιφέρειες και μετά τα κράτη και μόνο μετά έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση που βέβαια έχει να προσφέρει εργαλεία για τη δημιουργία τάσεων. Αλλά πρώτα πρέπει να χαράξουμε μια στρατηγική και εν συνεχεία να χωρίσουμε κάποιες αρμοδιότητες ούτως υπήν, ώστε οι περιοχές αυτές από τις οποίες φεύγει, τις οποίες εγκαταλείπει, πρέπει να μπορούν να αξιοποιήσουν αυτά τα κονδύλια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χούας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι λακωνικός γιατί με κάλυψαν οι προλαλήσαντες. Ε, πραγματικά είναι πολύ επίκαιρο αυτό το θέμα. Εγώ γνωρίζω πολύ καλά αυτό το θέμα γιατί κατάγομαι από μια περιοχή ε, που μοιάζει με, τα, αυτά που μας περιέγραψε η κυρία Ιράτσα ε, Γκαρσία γιατί ανήκουμε και εμείς στην Ιβηρική Χερσόνησο και από τις, από τις 308 δήμους που έχουμε 168 είναι αεροκατοικημένοι οπότε ενταμετωπίζουμε αυτό το φαινόμενο της απερίμωσης της υπαίθρου. Οπότε η πρώτη ευκαιρία που μπορεί να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να σταματήσει η απερίμωση, γιατί αυτή η απερίμωση δημιουργεί προβλήματα και στις αστικές ζώνες και στα αστικά κέντρα. Και πολλά από τα προβλήματα που ε, καλούμαστε να λύσουμε στις πόλεις είναι ακριβώς επειδή επιτρέψαμε αυτή τη μαζική απερίμωση και την ε, ενίσχυση της αστιφιλίας τα τελευταία χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν αφενός να, να αποφύγουμε την απερίμαση της υπαίθρου και ταυτόχρονα έτσι θα βοηθήσουμε την ελάφρυση των προβλημάτων των πόλεων. Ένα άλλο ζήτημα κέριο είναι το εξής. Έχουμε πολλές ε, δημόσιες επενδύσει ε, ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν χρειάζονται πια στην, στη, στην Ήπεθρο, γιατί έχουν απεριμωθεί οι περιοχές αυτές και έτσι όλες οι επενδύσεις που έγιναν στην υγεία, στην ε, ε, υδροδότηση, στην ηλεκτροδότηση, έχουν μείνει αχρησιμοποιητές, ανεκμετάλλευτες. Αυτό είναι μεγάλο κρίμα πραγματικά. Θα πρέπει όλα αυτά να τα σκεφτούμε όταν εξετάζουμε το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Επίσης θα πρέπει ταυτόχρονα να έχουμε και μια κατάλληλη πολιτική γεννητικότητας, γιατί δεν αρκεί μια τοπική πολιτική γεννητικότητας για να λύσουμε το πρόβλημα της γύρα του πληθυσμού. Χρειαζόμαστε πανευρωπαϊκή πολιτική. Επίση θα πρέπει να αποφύγουμε αυτή τη διχοτόμηση μεταξύ υπαίθρου και αστικών περιοχών. Γιατί ξέρουμε ότι το... Ε, και βραχυπρόθεσμα θα έχουμε ε, ε επίσης αύξηση τη αστιφιλίας, οπότε το το φαινόμενο της αποερήμωσης ε, θα ενισχυθεί, αλλά εγώ είμαι υπέρ των ε, πόλων ε, μέσων διαστάσεων, όχι των μεγάλων αστικών κέντρων. Και έτσι νομίζω θα επιτρέψουμε μεγαλύτερη παραμονή του πληθυσμού και στις, στην Υπέθρο. ώστε να μην έχουμε υπερμεγέθη αστικά κέντρα και να μην έχουμε ταυτόχρονα και απερίμωση της Ήπεθρου. Να μπορέσουν οι νέοι να παραμείνουν στους σε μικρότερους δήμους και κοινότητες. Πάντως, επαναλαμβάνω, είναι πολύ εύστοχη η πρόταση για αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας και θα συμβάλλω και εγώ στη διαμόρφωσή της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νίλσεν, έχετε το λόγο. Νομίζω ότι μπορώ να μιλήσω σου ειδικά, δεν είναι. Är det svenska? Jag kan prata Ωραία. Θα προσπαθήσω να τα καταφέρω στα αγγλικά λοιπόν αφού δεν μπορώ να μιλήσω σουηδικά. Θα σας πω δύο λόγια να απεικονίσω λίγο την κατάσταση στην ε, Σουηδία. Είχαμε και εμεί την ίδια συζήτηση γιατί τα προβλήματα είναι παρόμοια. Ναι, οι άνθρωποι που φεύγουν από την Ήπεθρο και που πηγαίνουν σε μεγάλε πόλει, αυτό συμβαίνει σε ολόκληρη την ε, Ευρώπη. Και οι ηλικιωμένοι ε, παραμένουν επιτόπου και σιγά σιγά περιμόνονται και πεθαίνουν κάποια ε, χωριά. Θα πρέπει ε, με κάποιο τρόπο να κάνουμε τις ε, περιφέρειες του Βορρά ε, να φαίνονται πιο ελκυστικές. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Με την εκπαίδευση. Με την εκπαίδευση. Θα πρέπει στις περιοχές αυτές να υπάρχει δυνατότητα έρευνας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πανεπιστημίων. Αυτή ήταν μια μεγάλη πολιτική μάχη που δώσαμε για να δημιουργήσουμε νέα πανεπιστήμια δεν το θέλαν αυτό οι συντηρητικοί γιατί λέγανε πρέπει να είναι μαζεμένα τα πανεπιστήμια όλα σε μία περιοχή αλλά έχουμε τώρα τρία πανεπιστήμια ε, στο βορρά της χώρας μου. Σε σχέση με τη χρήση δε των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων για την έρευνα, θα σας πω το εξής. Περίπου 80% ε, του, των κονδυλίων ε, του ορίζοντα 2020 ε, αφορούσαν ακριβώς μεγάλα πανεπιστήμια σε μεγάλες πόλεις, όχι μικρά πανεπιστήμια. Και αυτό είναι προβληματικό. Αυτό σημαίνει ότι στη Βόρεια Σουηδία το Περιφερειακό Ταμείο είναι πιο σημαντικό για τα πανεπιστήμια από ότι το πρόγραμμα Horizon 2020 γιατί μέσω των ε, περιφερειακών ταμείων ε, χρηματοδοτείται η έρευνα στα πανεπιστήμια αυτά. Αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε όμως είναι να αλλάξουμε τους κανόνες και του προγράμματος Horizon 2020 αλλά και άλλων προγραμμάτων έτσι ώστε όχι μονάχα τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια να παίρνουν τα ε, περισσότερα κονδύλια αλλά μέσω εδαφικών δικτών να τα παίρνουν και άλλα πανεπιστήμια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μόλκοβα. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα τα όσα είπε η συγγήτρια σε σχέση με την έκθεσή της και εκτιμώ ιδιαίτερο και την συζήτηση που λαμβάνει η χώρα ε, αυτή τη στιγμή γιατί το δημογραφικό πρόβλημα, η δημογραφική πρόκληση είναι μεγάλη όχι μόνο για συγκεκριμένες εδαφικές ενότητες αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, οι δημογραφικές αλλαγές είναι σημαντικές και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ας δούμε όμως και τι εργαλεία έχουμε ήδη στα χέρια μας. Δεν είναι και λίγα. Εάν θέλει κανείς να αλλάξει τις δημογραφικές ε, ε, τάσεις θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα είδος ομπρέλας που θα μπορούσε να βοηθήσει τους νέους δίνοντάς τους κάποια, κάποιο βαθμό ασφάλειας. Ε, είναι πολλοί αυτοί που θέλουν να ξεκινήσουν οικογένεια, να κάνουν παιδιά, αλλά εάν δεν έχουν ε, στέγη, αν δεν έχουν δουλειά, ε, προφανώς δεν ε, μπορούν να ξεκινήσουν ε, οικογένεια και ακόμα και αν έχουν στέγη, ακόμα και αν έχουν κάποια δουλειά, σε μικρές ε, πόλεις, σε μικρά χωριά δεν ξέρουν εάν θα μπορεί να βρουν κάποιον να τους βοηθήσει με τα παιδιά τους. Αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην έκθεση, γιατί εργαλεία υπάρχουν, αλλά θα πρέπει να είναι στοχευμένα, θα πρέπει να είναι συγκεκριμένα έτσι ώστε έτσι ώστε οι εκστρατείες πληροφόρησης ε, ε, να ξεπεράσουν πλέον ε, την προπαγάνδα για το πρόβλημα που μπορεί να αποτελέσει η μετανάστευση και άλλα ε, σχετικά. Θα πρέπει να γίνουν εκστρατείες ε, υπέρ της ασφάλειας, ε, να ξέρουν δηλαδή οι νέοι ότι μπορούν να βοηθηθούν στην οικοδόμηση του μέλλοντός τους. Σας λέω, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αρνούνται να κάνουν οικογένεια γιατί δεν ξέρουν αν θα μπορέσουν να τα καταφέρουν. Θα πρέπει να υπάρξουν οι απαραίτητες στεγαστικές πολιτικές ε, και ε, οπωσδήποτε να έχουμε και εκστρατείες πληροφόρησης σχετικά ε, με τη βοήθεια που μπορεί να δοθεί σε σχέση εκστρατείες επίσης όσον αφορά την αποσχόληση, όσον αφορά την δυνατότητα παροχής βοήθειας για μικρά παιδιά κτλ. Εάν μια γυναίκα αποφασίσει να μείνει στο σπίτι μέσω γονικής άδειας, τότε δεν έχει αρκετά χρήματα η οικογένεια. Ε, αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να το καταλάβουμε, γιατί συμβάλλει στις δημοκρατικές, συγγνώμη, δημογραφικές αλλαγές. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χάτμαν, έχετε το λόγο. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ε, και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτριά μας γιατί πραγματικά το θέμα είναι πολύ επίκαιρο και από τα πιο δύσκολα, τα πιο ακαθόδια, αλλά και τα πιο σπουδαία σοβαρά προβλήματα που θα αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί προλαλήσαντες μίλησαν για το θέμα αυτό. Εγώ ε, κατάγομαι από την Πολωνία ε, και κυρίως ε, μάλιστα από μια ανατολική περιοχή και το θέμα της απερίμωσης ε, μας προβληματίζει ιδιαίτερα γιατί μαστίζει ιδιαίτερα την Ανατολική Πολωνία από όπου και κατάγομαι. Ε, κατά τη γνώμη μου, ένα από τα πιο σημαντικά θέματα είναι αυτά ε, της ε, γύρας του πληθυσμού και της αντιμετώπιση της απερίμωσης. Βέβαια, στην πρώτη γραμμή του πυρός ε, για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος είναι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι δήμοι, οι κοινότητες και μετά οι πόλεις. Νομίζω όμως ότι η καλύτερη ευρωπαϊκή πολιτική, ενωσιακή πολιτική που μπορούμε να έχουμε στον τομέα αυτό, δεν θα βοηθήσει αν δεν εμπλέξουμε ενεργά τους τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες, ε, τους δήμους και κοινότητες ε, και τις πόλεις. Γιατί οι τοπικοί και περιφερειακοί φορείς είναι σε καλύτερη θέση και γνωρίζουν τι ακριβώς πρέπει να κάνουν, αλλά τους λείπουν τα εφόδια, τους λείπουν τα μέσα. Θα πρέπει λοιπόν εμεί να του βοηθήσουμε, γιατί αυτοί είναι σε στην κατάλληλη θέση να λύσουν το πρόβλημα. Αλλά χρειάζονται, παραλαμβάνω, του μηχανισμού, τα μέσα και τα εργαλεία. Οπότε επανερχόμαστε εδώ σε ένα παλιότερο πρόβλημα, σε ένα πρόβλημα που μας απασχολεί εδώ και χρόνια ολόκληρα και αφορά την πολιτική συνοχή και την ελαστικότητα, την ευελιξία της πολιτικής συνοχής. Εδώ θα ήθελα να προσυπογράψω και να ενισχύσω τη θέση του κυρίου Λάμπερτ ότι δεν χρειαζόμαστε ένα ακόμη ταμείο για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Δεν χρειάζεται για κάθε νέο πρόβλημα που έχουμε να επινοούμε και ένα νέο ταμείο. Αρκεί να φροντίσουμε ε, να εξασφαλίσουμε συμπληρωματικότητα και συντονισμό μεταξύ των μηχανισμών και των εργαλείων που έχουμε και των ταμείων. Και παραλαμβάνω να εμπλέξουμε ενεργά τους τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες, ιδιαίτερα αυτούς που μαστίζονται ιδιαίτερα από το πρόβλημα. Και ό,τι κάνουμε θα πρέπει να είναι καινοτόμο, νεοτεριστικό βέβαια. Αλλά δεν πρέπει να χρηματοδοτούμε μόνο ε, καινοτόμα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί εδώ το πρώτο ουσιώδη στοιχείο ε, του προβλήματος για να μπορέσουν ο κόσμος, να μπορέσει ο κόσμος να βρει προοπτική και ελπίδα για να παραμείνει στο χώρο είναι να ενισχύσουμε τις υπηρεσίες παιδείας, ε, υγείας, τα είπαν οι δεν χρειάζεται να παραλάβω κι εγώ. Μόνο έτσι, ενισχύοντας ε, την κατάσταση αυτή και βελτιώνοντας ε, την κατάσταση, θα παραμείνει ο κόσμος στην Ήπεθρο. Και επαναλαμβάνω να ενισχύσουμε τη συμπληρωματικότητα και το συντονισμό των ταμείων που ήδη έχουμε. Του Κοινωνικού Ταμείου, του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ε, επίσης έχουμε και την κοινή γεωργική πολιτική και στον τομέα αυτό φέρει μεγάλη ευθύνη η κοινή γεωργική πολιτική. Θα πρέπει λοιπόν και στις συζητήσεις που θα κάνουμε για το τι μέλη γενέστε μετά το 2020 λοιπόν, δηλαδή 20, να δούμε που έγκυται τα βασικότερα προβλήματα και να βρούμε την συμπληρωματικότητα μεταξύ της ε, πολιτικής συνοχής και της κοινή γεωργικής πολιτικής. Μόνο με συμπληρωματικότητα, με καλύτερο συντονισμό των μηχανισμών, αλλά πρώτα απ' όλα ε, με μεγαλύτερη ελαστικότητα και ευελιξία απέναντι στους δικαιούχους των ταμείων. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να βοηθήσουμε πραγματικά όσους ε, ασχολούνται με το πρόβλημα αυτό στο, στην πρώτη βαθμίδα, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Και νομίζω ότι με τέτοια συμπληρωματικότητα, συντονισμό και συνεργασία θα λύσουμε και πολλά προβλήματα. Ευχαριστώ κυρία Μπρέσο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την συνάδελφο γιατί όπως φαίνεται και από τη συζήτηση ε, αναφέρθηκε σε ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους γιατί όλοι έχουμε θυγεί, έχουμε πληγεί από αυτά τα δύο σκέλη του δημογραφικού ε, προβλήματος. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να ξεχωρίσουμε τα δύο ζητήματα. Έχουμε ζήτημα γύρανσης γενικευμένο του πληθυσμού και στις αστικές περιοχές και παντού στην Ευρώπη και για να αντιμετωπιστεί χρειάζεται συντονισμός των ε, πολιτικών, των κοινωνικών για την οικογένεια ε, έτσι ώστε να μπορέσει ο κόσμος ε, να ξεφύγει από τη φτώχεια, μια πολιτική συγκεκριμένη για τις γυναίκες, δηλαδή ένα σύμπλεγμα πολιτικών οι οποίες θα αναπτύσσονται και θα συντονίζονται καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειάζεται λοιπόν να ανεληφθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες έτσι ώστε ε, να ε, αποφασίζουν οι οικογένειες να κάνουν περισσότερα παιδιά ε, γιατί ξέρουμε ότι τα λίγα παιδιά είναι απόρρια των προβλημάτων των κοινωνικών, της φτώχειας και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Τώρα έχουμε το άλλο πρόβλημα ε, που αφορά την μείωση της πυκνότητας του πληθυσμού σε συγκεκριμένες περιοχές. Γιατί δεν ισχύει παντού αυτή η μείωση σε κάποιες ορεινές ε, περιοχές της Άλπης ας πούμε υπάρχουν ε, πάρα πολλές ε, περιφέρειες, πολλά, πολλά μέρη όπου σταμάτησε η μείωση του πληθυσμού και μάλιστα έχει ξεκινήσει και διαδικασία επιστροφής στην Ήπεθρο ή στις ορεινές περιοχές. Υπάρχουν όμως άλλες περιοχές όπου η μείωση είναι διαρκής. Τώρα, ε, ε, εκεί ακριβώς ε, θα πρέπει να δράσουν τα διαρθωτικά ταμεία θα πρέπει τα διορθωτικά ταμεία να κατανοήσουν ακόμα περισσότερο ότι ε, πρέπει να διαφοροποιηθούν οι πολιτικές. Ε, από τη μία πλευρά έχουμε τις πολιτικές οι οποίες θα ενδυναμώσουν την οικονομία κτλ. Από την άλλη όμως έχουμε ε, την προσπάθεια να αποκτήσουν ίδιο ρόλο οι περιφέρειες. Εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να λυθεί μέσω μακροοικονομικών οικονομικής αιρεσιμότητας πολύ συχνά ε, τα κράτη, οι περιφέρειες επενδύουν κονδύλια ε, για την ανάπτυξη ε, περιοχών ε, με ε, μικρή πυκνότητα ε, πληθυσμού και ταυτόχρονα όμως από την άλλη πλευρά αφαιρούν υπηρεσίες οι οποίες είναι απαραίτητες έτσι ώστε να μπορέσουν αυτοί οι πληθυσμοί να παραμείνουν σε αυτές τις περιφέρειες γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να παραμείνουν οι άνθρωποι αυτοί σε αυτές τις περιοχές εάν δεν έχουν κανονική ανάπτυξη και αν δεν έχουν και την παροχή των ελάχιστων υπηρεσιών. Εγώ λοιπόν προτείνω να ε, μην λησμονούμε ακριβώς αυτό, δηλαδή ότι όσον αφορά τις δημόσιες και οι ιδιωτικές υπηρεσίες ε, στις περιφέρειες με μικρή πυκνότητα πληθυσμού, ότι ε, δεν μπορούμε να αφήσουμε στα χέρια της αγοράς την διατήρηση των υπηρεσιών. Ε, σε πολλές ε, περιπτώσεις ε, οι μικρές κοινότητες αντιμετωπίζουν ακόμα περισσότερα οικονομικά προβλήματα. Επομένως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και αυτό το πρόβλημα διασφαλίζοντας ότι μέσα από δημόσιες συνεισφορές θα υπάρξει η, θα υπάρξει η παροχή δημοσίων και ιδιωτικών υπηρεσιών έτσι ώστε να μπορέσει να κρατηθεί ο πληθυσμός σε αυτές τις περιφέρειες. Υπάρχουν και άλλες πολιτικές οι οποίες είναι επιτυχείς, όπως είναι ας πούμε ε, η ονομασία των προϊόντων ή όπως είναι οι εναλλακτικέ μορφές ενέργειας. ενέργειας. Ε, είναι πολλές ε, οι περιπτώσεις όπου ξεπεράστηκαν προβλήματα μέσα από αυτές τις πολιτικές που ανέφερα προηγουμένως αλλά εμείς λέμε ότι ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να διασφαλιστεί ένα καλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών ε, σε, αυτήν, σε αυτές τις περιφέρειες. Και όταν λέω αναφέρομαι σε υπηρεσίες δεν αναφέρομαι μονάχα στο ταχυδρομείο ας πούμε γιατί σε, μια μικρή, σε ένα μικρό χωριό μπορεί ε, το ταχυδρομείο να είναι σε ένα άλλο μαγαζί. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Αναφέρομαι σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, σε πολιτικές ε, αρρωγής, ε, εκεί όπου η αγορά δεν έχει καλύψει τα κενά, ε, να υπάρχει πάντα η δυνατότητα κρατικών επιδοτήσεων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Αυτά ήταν τα σχόλια της, Επιτροπή, της Επιτροπής μας. Θα δώσω τώρα το λόγο στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Χαπάκα. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και την εισηγήτρια που επισήμανε αυτό το εύστοχο και επίκαιρο θέμα. Και μάλιστα ειδικά φέτος που εξετάζουμε την ε, τρέχουσα πολιτική, την εφαρμογή της και τις μελλοντικές προοπτικές. Και μάλιστα επισημάνεται πολλά ζητήματα που συνδέονται με αυτές τις προκλήσεις και αυτό το θέμα και όχι μόνο την πολιτική συνοχής. Έχουμε πολλά μέσα ε, και ταμεία που μας βοηθούν να αντιμετωπίσουμε το θέμα και στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού υπάρχουν δυνατότητες για καλό συντονισμό μεταξύ τους και υπάρχουν πολλές δυνατότητες για τη χρήση, αξιοποίηση αυτών των κονδυλίων και σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο ώστε να είμαστε όσο πιο κοντά γίνεται στην εμφάνιση των προβλημάτων. Οπότε προσβλέπουμε και σε στη συνεργασία για το θέμα αυτό και στη συζήτηση για μετά το 2020 και το Φόρουμ της Συνοχής και η Έκθεση της Συνοχής θα μας δώσουν το πλαίσιο και την ευκαιρία να συζητήσουμε και να αναλύσουμε τις μελλοντικέ προοπτικές. Σας ευχαριστώ κυρία Πέρες. Θέλετε να ολοκληρώσετε παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, για τις παρατηρήσεις τους. Νομίζω ότι ήταν πολύ καρποφόρα συζήτηση και ήταν η πρώτη ανταλλαγή απόψεων ε, με κατάθεση όμως πολύ εύστοχων ε, και σημαντικών προτάσεων. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι η κατάσταση είναι ανησυχητική, θα πρέπει να εγγύψουμε σε αυτήν και να αναζητήσουμε τρόπους είτε σε θεσμικό επίπεδο από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα είτε σε άλλο επίπεδο για να διορθώσουμε την κατάσταση. Αναφέρθηκε και η αρχή της επικουρικότητας. Συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση αυτή, γιατί οι τοπικές και περιφερειακές αρχές νιώθουν στο πεζί τους αυτές τις πιέσεις και αντιμετωπίζουν από κοντά αυτή την πραγματικότητα. Θα πρέπει λοιπόν να τους εφοδιάσουμε με μέσα και εργαλεία ώστε να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες τους και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά αυτή την πραγματικότητα που είναι περίπλοκη, πολυσύνθετη γιατί όλοι συμφωνούμε ότι δεν θα επιλύσουμε την κατάσταση με ένα μαγικό ραβδάκι ούτε υπάρχει μία ενιαία και μοναδική λύση για να αντιμετωπίσουμε όλες τις δημογραφικές προκλήσεις. Τώρα, για το αν θα χρειαζόμαστε και ένα ειδικό ταμείο γι' αυτό και αυτό το ζήτημα ε, είναι συζητήσιμο. Θα δούμε ποια είναι η κρατούσα άποψη περί κατά ενός νέου ταμείου. Πάντως θα πρέπει να δούμε πρώτα πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα υφιστάμενα μέσα και εργαλεία που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της απερίμωσης, της εγκατάλειψης της υπαίθρου. Γιατί ακούμε τους ε, τοπικούς και περιφερειακούς φορείς ε, που λένε ότι δεν ε, φτάνουν ε, τα κονδύλια, τα ευρωπαϊκά κονδύλια στην Ήπεθρο για να κρατήσουν τον πληθυσμό εκεί και να αποφύγουν την αστιφιλία. Το θέμα δεν είναι ότι θα επιρρύψουμε ευθύνε στην Α ή Β διοίκηση τοπική περιφερειακή, αλλά κάτι συμβαίνει και τα ευρωπαϊκά κονδύλια δεν φτάνουν ε, με αποτελεσματικό τρόπο στην Ήπεθρο ώστε να παραμείνει ο πληθυσμό ε, σε αυτό το επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε έναν καλό προγραμματισμό των πολιτικών ώστε να καταφέρουμε να επιλύσουμε ε, αυτά τα προβλήματα. Μίλησαμε για πολιτικές ε, συνδυασμού του επαγγελματικού προσωπικού βίου, της ενίσχυσης της γεννητικότητας. Θα πρέπει να συντονίσουμε τις προτάσεις μας και τις δράσεις μας αυτή την εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει στον κοινωνικό πυλώνα τα θέματα τα συναφή με τη, το συνδυασμό, τη συμφιλίωση προσωπικού και επαγγελματικού βίου. Επίσης θα πρέπει να δώσουμε ευκαιρία στα νέα ζευγάρια να μπορούν να αποφασίζουν πού θα διαβιώσουν. Δεν θα υποχρεώσουμε κανένα να παραμείνει στην Ήπεθρο, απλώς θα δώσουμε ελευθερία επιλογής σε όσους ε, θέλουν, σε όσους επιθυμούν να παραμείνουν στα χωριά τους, ε, στη γενέτειρά τους, να έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Γιατί μερικές φορές εξαναγκάζονται σε έξοδο, σε μετανάστευση, γιατί ακριβώς ε, δεν έχουν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο τις υποδομές μεταφορών, παιδείας, υγείας και τις υπηρεσίες που αναφέραμε. Επίσης θα πρέπει να κάνουμε ένα καλό προγραμματισμό και μάλιστα έξυπνο προγραμματισμό. Γιατί δεν λέμε ότι θα πρέπει όλοι οι Δήμοι να έχουν κέντρο υγείας, εκπαιδευτικό κέντρο, κέντρα αναψυχής ε, ή αθλητισμού. Θα πρέπει να κάνουμε τον καλύτερο προγραμματισμό ώστε όσοι διαμένουν στην Ήπεθρο να έχουν πρόσβαση σε όλες τις σχετικές υπηρεσίες. Και θα πρέπει να συμβάλλουμε όλοι στη συζήτηση αυτή που είμαι σίγουρη ότι θα είναι πλούσια και καρποφόρα και ελπίζω να καταλήξουμε σε προτάσεις ε, ώστε να μας, που θα μας επιτρέψουν να κρατήσουμε τον πληθυσμό στην Ήπεθρο για να αναχαιτήσουμε όλες αυτές τις επικίνδυνες τροπές που επισημάναμε. Και ήδη από την επόμενη εβδομάδα θα υποβάλω ένα σχέδιο ε, εγγράφου για να αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω συζήτηση και χάρη και στις δικές σας παρατηρήσεις πιστεύω θα καταλήξουμε σε μια έκθεση που θα προσφέρει λύσεις σε ένα κοινό μας μέλημα και που είναι η αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων και της απώλειας πληθυσμού. Ευχαριστώ. Θα περιμένουμε τον Ιούνιο την έκθεσή σας και θα συνεχίσουμε τότε τη συζήτηση. Οπότε τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο της μέρης που είναι ανταλλαγή απόψεων ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ε, εξελίξεις σε σχέση με το αστικό θεματολόγιο. Δεν χρειάζεται καν να σα πενθυμίσω πόσο πολύ ε, προσπάθεια έχει επενδυθεί σε ό,τι το σύμφωνο του Άμστερνταμ και το αστικό θεματολόγιο. Ε, μάλιστα η Επιτροπή μας κατάρτισε ειδική έκθεση και συμμετείχε, ε, είχαμε ενεργά σε όλε τι εκδηλώσει από εκείνου με την Επιτροπή των Περιφερειών και την Επιτροπή Κοτέρ της Επιτροπής των Περιφερειών τον Ιούλιο θα ξαναγίνει συνάντηση με την Επιτροπή ΚΟΤΕΡ τη Επιτροπή των Περιφερειών για το θέμα αυτό. Το επίκεντρο ταστικό θεματολογίο για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι η ε, δημιουργία 12 εταιρικών σχέσεων. Και τα σχέδια δράση για τι εταιρικέ αυτέ σχέσει είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και εστιάζουν τι προσπάθειε των διαφόρων θεσμικών οργάνων στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αστικές περιοχές ως προς την ανάπτυξη. Μέχρι τα τέλη του έτους ε, περιμένουμε έκθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το Συμβούλιο με θέμα το πώς προχωρά το αστικό θεματολόγιο και πώς προχωρούν και αυτές οι εταιρικές σχέσεις και βέβαια και εμείς θα έχουμε τις δικές μας ε, συνεδριάσεις, τις δικές μας συναντήσεις και σήμερα θέλουμε να ενημερώσουμε τα μέλη της Επιτροπής. Ο κύριος Πόπενς είναι εδώ αναπληρωτής Γενικό Διευθυντής της ΓΔ ΡΕΓΚΙΟ. Χαίρομαι που τον έχουμε κοντά μας ε, και θα τον παρακαλέσω να μας κάνει μια εισαγωγή. Στο θέμα αυτό, που είναι και βάση τη συζήτησή μας. Μετά από την εισαγωγή αυτή θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε την εισαγωγή του κ. Πόπης. Παρακαλώ το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, Θέλω να εκφράσω ευχαριστήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όλων όσων συμμετείχαν ε, στην εκπόνηση του αστικού θεματολογίου και την Επιτροπή Ρέτζι που μας παρήχε ζωτική υποστήριξη. Ιδίω δε εν καιρό κρίσης, μα μην ε, διαφορετικών κρίσεων και ε, ευάλωτων καταστάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το σύμφωνο το Άμστερνταμ και το σχέδιο το οποίο δρομολογήθηκε δείχνει πώς μπορούν να συνεργαστούν τελικά ε, αποτελεσματικά στο εσωτερικό σχέσεων διάφοροι φορείς. Και η βασική ορολογία στο αστικό θεματολόγιο περιλαμβάνει τον όρο συνεργασία βέβαια. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε προχωρήσει και εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορώ να σας ε, διαβεβαιώσω ότι πάρα πολύ ενεργά εργαζόμαστε στο πλαίσιο του αστικού θεματολογίου για να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατόν. Είναι προφανές ότι αυτό είναι σημαντικό δεδομένων των προβλημάτων αλλά και των προκλήσεων και ευκαιριών όμως που υπάρχουν, εξακολουθούν να υπάρχουν στις αστικές περιοχές που είναι κοντά στους πολίτες. Αντιμετωπίζοντας λοιπόν τα προβλήματα και τις προκλήσεις ε, κάνουμε πράγματα που είναι πάρα πολύ ε, που ενδιαφέρουν πάρα πολύ του πολίτε. Είπατε ότι υπάρχουν αυτά τα σχέδια συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών Ευρωπαϊκή Επιτροπή πόλεων και άλλων πληκωμένων φορών, ΜΚΟ. Συμμετέχει βέβαια και το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή των Περιφερειών. Αυτή είναι η προσέγγιση που ακολουθήσαμε στην κατάρτιση αυτών των εταιρικών σχέσεων. Σε κάθε εταιρική σχέση επικεφαλή είναι ένα εκ των φορέων που είναι τελείω διαφορετική. Παραδείγματο χάρη στην εταιρική σχέση για τη μετανάστευση έχουμε την ΓΔ Home από την Κομισιόν, αλλά σε άλλε περιπτώσει ε, ηγούνται των ε, εταιρικών σχέσεων κάποιε πόλει ε, ή κάποια κρατημέλη. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση για συμπερίληψη στι εταιρικέ σχέσει. Εκδηλώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον από διάφορου φορεί. Και όπω γνωρίζετε, προχωρήσαμε με τι τέσσερι πρώτε εταιρικέ σχέσεις που ήταν ε, αστική περιουσία, μετανάστευση, ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα και ε, στέγαση, οξέα προβλήματα, μεγάλες προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν. Σε αυτές τις εταιρικές σχέσεις περιμένουμε τα σχέδια δράση είναι έτοιμα μέχρι το καλοκαίρι, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία διαβούλευσης, δημόσια διαβούλευση στις ιστοσελίδες μας ήδη από Αύγουστο Ιούλιο και μπορούμε να έχουμε μια συζήτηση έτσι με τις πόλεις ε, και τα κρατημέλη από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ήδη. Στα σχέδια δράση τρία είναι τα βασικά σημεία που θα να άξονα χρηματοδότηση, γνώση και νομοθεσία. Προσπαθούμε λοιπόν όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένα να αντιμετωπίσουμε τους τρεις αυτούς βασικούς τομείς, διότι είναι προφανές ότι αυτό που ε, κάνουμε με την νομοθεσία μας επηρεάζει και δεν μιλάμε μόνο για την ευρωπαϊκή αλλά και για την εθνική νομοθεσία η οποία επηρεάζει. Παραδείγματο την ποιότητα του αέρα, τη μετανάστευση, πώς αντιμετωπίζουν τα θέματα αυτά οι πόλει. Η χρηματοδότηση επίση είναι πάρα πολύ σημαντική. Υπάρχουν διαφορετικέ πηγέ χρηματοδότηση για τις πόλεις, αλλά ενίοτε πρέπει να δούμε πού υπάρχουν κενά και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε και να στοχεύσουμε καλύτερα, καθοδηγήσουμε τις πόλεις ώστε να αναζητήσουν και να βρουν τη σωστή χρηματοδότηση. Και βέβαια η ανταλλαγή γνώσεων είναι κάτι που δεν πρέπει να υποτιμηθεί σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν συγκρίνουμε τις διάφορες ε, περιοχές της Ευρώπης και τις διάφορες πόλεις. Ε, υπάρχει ανάγκη λοιπόν ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και ε, ανταλλαγή καλών παραδειγμάτων και γνώσεων. Δηλαδή πολλές φορές δεν γνωρίζουν οι πόλεις, οι δήμοι, τι πρέπει να κάνουν. Πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε διάφορα μέσα στην ανταλλαγή αυτών των βέλτιστων πρακτικών. Μια από τις βασικές ε, γραμμές της Κομισιόν ήταν ο εξορθολογισμός της εργασίας μας. Είδαμε ότι πολλές τομεακές πολιτικές επηρεάζουν τις αστικές περιοχές που Μόνο αν εφαρμοστούν σωστά μπορούμε να πετύχουμε. Προσπαθούμε πραγματικά να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας, συντονίσει τρένη γάμα δελτα ρέγγιο, αλλά και άλλες γενικές διευθύνσεις συμμετέχουν σε συγκεκριμένες εταιρικέ ε, σχέσεις, όπως είναι η ψηφιακή οικονομία, για παράδειγμα. Υπάρχει λοιπόν εσωτερική κινητοποίηση και ε, εντό κομψιών με του διάφορου γιατί πρέπει να πω ότι έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα και βάσει αυτών θα κρίνουμε και τα ε, σχέδια δράσης και την αποτελεσματικότητά τους. Ο στόχο μα είναι κάποιε πιο κοινέ έννοιε, κοινά κόνσεπτ για το μέλλον. Έχουμε την έννοια των εφιών πόλεων, υπάρχουν διάφορα μέσα. Αλλά αυτό που θέλουμε να προωθήσουμε στη ΓΔ Ρέγγιο είναι κάτι πιο ομοιόμορφο και αναρμονισμένο. Επίση, ε, κάνουμε και τις ε, μελέτες εδαφικού αντικτύπου. Ένα πολύ μεγάλο αίτημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα ε, σε εξέλιξη στην Γαμματελτα Ρέγγιο και δεν ασχολούμαστε βέβαια μόνο με τις αστικές πρίξεις αλλά και με την Ήπεθρο. Θέλουμε λοιπόν αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα να το προχωρήσουμε. Έχει άλλωστε αναπτύξει η Επιτροπή των Περιφερειών μια σημαντική μεθοδολογία. Συνεργαζόμαστε στενά με την Επιτροπή των Περιφερειών. Στόχος με αυτά τα πιλωτικά προγράμματα είναι να δούμε πώς μπορούμε αυτήν την ε, μεθοδολογία να την εντάξουμε στις ε, μελέτες αντικτύπου, την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Όπως είπα, αυτό που πρέπει να γίνει, γιατί αυτή είμαστε στη μέση, αν θέλετε, έκανα τον απολογισμό, σας είπα που βρισκόμαστε, τώρα επεξεργαζόμαστε αυτή την έκθεση προς το Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά τι εταιρικέ σχέσει, ε, το θα έχουμε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο τα πρώτα παραδοτή αποτελέσματα και θα προχωρήσουμε μετά και τις επόμενες εταιρικές σχέσεις. Στην Περατισλάβα είχαμε την κυκλική οικονομία, την κινητικότητα, τις δεξιότητες ε, και περιμένουμε εκεί γύρω στις αρχές του 2018 να έχουμε σχέδια δράσης. Το θέμα είναι να δείξουμε τι συγκεκριμένες δράσεις προτείνονται και θα υπάρξουν δράσεις για τα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης ως Κομισιόν φυσικά θα δούμε πολύ σοβαρά τι μπορούμε εμείς να κάνουμε, αλλά δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι πρόκειται για εταιρική σχέση. Υπάρχει χώρο συζήτησης για να δούμε οι πόλεις, ε, οι ΜΚΟ, οι Δήμοι, τι κάνουν, πώς μπορούν να συνεισφέρουν. Ο μεγάλος είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επίσης, για το συντονισμό και για την ε, οργάνωση της συζήτησης. Προσπαθούμε επίσης ε, σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα πληροφοριών να την εξορθολογήσουμε. Θέλουμε να έχουμε μια νέα θηρίδα, έχουμε την, στην ιστοσελίδα μας ε, τη σχετική, το σχετικό χώρο που μπορούν όλοι να δουν ε, τα προγράμματα, τις εταιρικές σχέσεις. Και με την ΕΤΕΠ προσπαθούμε με αυτή την νέα θηρίδα να έχουμε ε, συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα μπορέσουν να βοηθήσουν τους φορείς, να υπάρχει μια στοχευμένη βοήθεια λοιπόν στις, ε, στις πόλεις, να έχουν την καθοδήγηση, ε, να αναπτυχθούν σωστά ολοκληρωμένες αναπτυξίες στρατηγικές και επίσης ε, πρόσβαση στη χρηματοδότηση, να εξασφαλιστεί. Η χρηματοδότηση υπάρχει, αλλά οι πόλεις κάποιες φορές τελούν υποσύγχυση, ως προς το που να βρουν την κατάλληλη πηγή χρηματοδότηση. Πρέπει να βοηθήσουμε λοιπόν και πρέπει να ακούσουμε τις πόλεις. Έχουμε 10 πόλεις ε, στο focus group. Στόχος μας είναι να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις πραγματικές ανάγκες των πόλεων, να μην κάνουμε κάτι γενικό δηλαδή. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να δούμε τι γίνεται εντός της πολιτικής συνοχής και εντός των προγραμμάτων που εκτελούμε. Έχουμε μια μελέτη και έχουμε και εσωτερικό που θα λαμβάνει το Σεπτέμβριο. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι πέραν της ΕΤΕΠΑ που έχει το δικό τους ε, σύστημα, τα δόνια, έχουμε τις τράπεζες, υπάρχει και πολύ μεγάλη χρηματοδότηση που προβλέπεται για τις πόλεις. Ε, έχουμε το άρθρο 7 του ΕΤΕ ότι θα πρέπει, του ΕΤΠΑ που λέει ότι θα ε, υπάρχουν συγκεκριμένα ποσοστά χρηματοδότηση. τους χάρη 10% προβλέπει το άρθρο 7 για τις πόλεις απευθείας. Τα κράτη-μέλη έχουν δεχθεί την ιδέα αυτή. Βέβαια, τον τελικό λόγο για την επιλογή των σχεδίων τον έχουν οι πόλει. Θέλουμε να δούμε επίση πώ μπορούμε να προχωρήσουμε σε απλούστευση, να μην υπάρχει υπερβολικό διοικητικό φόρτο, έλεγχη, αλλά να μπορούν να εστιάσουν την προσοχή του οι πόλει στην επιλογή των κατάλληλων σχεδίων. Έχουμε επίση την ολοκληρωμένη στρατηγική. Αυτή είναι και η προπόθεση. Βοήθησε πολλέ πόλει να κατανοήσουν προ τα που πρέπει να κατευθυνθούν και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις με ολιστικό τρόπο. Γνωρίζουμε όλοι ότι είναι μοχλή οικονομική ανάπτυξη οι πόλη, αλλά ε, σωρεύουν και προβλήματα. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση είναι πολύ χρήσιμη αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας και βλέπουμε με ικανοποίηση ότι λειτουργεί σωστά. Επίσης υπάρχουν εδαφικά εργαλεία ITIs κτλ. Χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή του άρθρου 7. Υπάρχουν λεγόμενες λειτουργικές, τα λειτουργικά εδάφη, περιφέρειες, δεν μιλάμε μόνο για πόλεις δηλαδή. Εστιάζουμε συνεργασία μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών. Αυτό πρέπει να το αναπτύξουμε περαιτέρω. Όλο και περισσότερα είναι τα στοιχεία που θα έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι το Σεπτέμβριο. Και πάνω σε αυτά θα οικοδομήσουμε τι προσπάθειέ μα. Με βάση όμω τα στοιχεία που έχουμε ήδη στη διάθεσή μα, αυτά τα εδαφικά εργαλεία έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερω χρήσιμα. Τα έχουν χρησιμοποιήσει διάφοροι φορεί για την αντιμετώπιση των εδαφικών προκλήσεων. Αν δε τα σχετίσουμε και με τη σωστή θεματική συγκέντρωση, στο μέλλον μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε επιτόπου τι ανάγκε. Γιατί δηλαδή, φυσικά ανάλογα με την περιφέρεια και ανάλογα με το έθνο είναι διαφορετικέ οι ανάγκε. Υπάρχουν εδάφη και περιοχές με συγκεκριμένες γεωγραφικές ανισότητες και ανισορροπίες, όπως είναι οι νησιωτικές περιοχές, οι ορεινές περιοχές. Με αυτά τα ETIs αναπτύσσουμε μια ανταυτική προσέγγιση που βασίζεται στη συνεργασία αστικών αγροτικών περιοχών. Πρέπει να δώσουμε ευκαιρία σε αυτές τις περιοχές να αντιμετωπίσουν τα ιδιαίτερα τους προβλήματα. Η δουλειά συνεχίζεται όπως βλέπετε. Έχουμε και κάποιες καινοτόμες αστικές δράσεις, ένα πολύ ενδιαφέρον εργαλείο. Είναι η πρώτη φορά που το εφαρμόζει το μέσο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είχαμε μια δεύτερη προκήρυξη. Ε, στην πρώτη υπάσκηση υποβολή ε, προσφορά είχαμε 400 αιτήσει από πόλει απευθεία. Για μετανάστευση, ενέργεια και πολλού άλλου τομεί. Και είναι ενδιαφέρον. Δυστυχώ μόνο 18 ε, τέτοια σχέδια μπορέσαμε να τα εγκρίνουμε Υπάρχει τεράστια ζήτηση για στρατηγικά σχέδια και θέλουμε να βελτιώσουμε. Για τη δεύτερη, προς το δεύτερη προκήρυξη είχαμε 200 σχέδια. Θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε λοιπόν να διοχετεύσουμε τα κονδύλια. Είναι επιτυχημένη η προσπάθεια και στο Steering Committee το είπαμε. Δεν περιμέναμε καν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως είπα λοιπόν, θα έχουμε μέχρι τα τέλη του έτους την έκθεση προς το Συμβούλιο. Πρέπει να δούμε πρώτα τα συγκεκριμένα σχέδια δράση, τι προτινόμενε δράσει, να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία στα χέρια μα. Περιμένουμε να έχουμε συγκεκριμένε προτάσει. Μετά θα πρέπει να αναλύσουμε την συμπέριψη στα προγράμματα, πάντα μέχρι τα τέλη του έτου και έπειτα επειδή υποστηρίζουμε το βασικό θεματολόγιο, ε, θα δούμε και σφαιρετέρω διασυνδέσεις αστικού και αγροτικού επίπεδου και θα οργανώσουμε στο Ρότερνταμ ένα φόρουμ πόλεων για να βγούμε λίγο από τις Βρυξέλλες. 27 και 28 Νοεμβρίου. Τρεις μέρες λέει ο Και ελπίζω να συμμετάσχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα είναι πάρα πολύ πολύτιμη η δική σα συμμετοχή. Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια εποχή που το μέλλον της Ένωσης ε, είναι υποσυζήτηση και ιδίως τα οικονομικά, χρηματοοικονομικά ζητήματα. Όπου πάω βλέπω πόσο μεγάλη ζήτηση υπάρχει για την πρόθεση του αστικού θεματολογίου, αλλά όχι μόνο, και αυτή τη αδαφική προσέγγιση εν γέννη. Στη Μάλτα τα συζητήσαμε προς Χτες και η Προεδρία εξεργάζεται εντατικά ε, ένα πρόγραμμα ε, για τα εδαφικά ζητήματα. Νομίζω λοιπόν ότι είναι καλό ο καιρό, καλή στη χρονική στιγμή να τα συζητήσουμε, να δούμε τι στοιχεία έχουμε στη διάθεσή μα και τι μπορούμε να κάνουμε και στο μέλλον. Σα ευχαριστώ και πάλι που με καλέστε και βέβαια είμαι στη διάθεσή σα να απαντήσω τι ενδεχόμενε ερωτήσει και όπω είπα αργότερα φέτο θα σας δώσουμε περισσότερα στοιχεία, γραφήματα, νούμερα γιατί προς το παρόν η δουλειά είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ευχαριστώ. Thank you very much. Thank you for this information. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος, για τις ε, πληροφορίες που μας δώσετε και βεβαίω θα παρακολουθήσουμε την πρόοδο και θα ξαναέρθουμε σε επαφή και πριν από το τέλος του χρόνου ε, για την ε, κοινή μα συνάντηση με την Επιτροπή Κοτέρ. Η κυρία Βέστβαλ έχει πρώτο λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ε, έκθεση που μας ε, κάνατε, έτσι ώστε να δούμε πώς έχουν τα πράγματα όσον αφορά το αστικό θεματολόγιο. Ε, νομίζω ότι ψηφίσαμε μια καλή έκθεση όχι μόνο εδώ στην Επιτροπή μας, ε, αλλά και στην Ολομέλεια. Και είπαμε με πολύ ε, καθαρό και ξεκάθαρο τρόπο ε, ότι ορισμένα πράγματα είναι πολύ σημαντικά. Θα επανέλθω σε αυτά τα οποία είπαμε όσον αφορά το δημογραφικό πρόβλημα για να τονίσω ότι είναι μεγάλος ο δεσμός ανάμεσα στις αστικές και μη αστικές περιοχές και πόσο σημαντικός είναι ο, δεσμός ανάμεσα στην Ήπεθρο και την, ε, τις αστικές περιφέρειες και πώς αυτός ο δεσμός πολλές φορές είναι αρνητικός. Ε, ή αναφέρατε κι εσείς τον ρόλο του Κοινοβουλίου και υπογραμμίσατε τη σημασία του ρόλου αυτού, όχι μονάχα στην αρχή, στο ξεκίνημα των διαδικασιών, αλλά και στο τέλος. Ε, γι' αυτό σας παρακαλώ, όποτε έχετε στη διάθεσή σας ε, συγκεκριμένα στοιχεία, να μας τα δώσετε. Είπατε κι εσείς ε, ότι η συνοχή ε, είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό, βρίσκεται πρώτων πυλών τα στοιχεία της επόμενης, ε, της μελλοντικής, μάλλον στην επόμενη μελλοντική πολιτική συνοχής, το αστικό θυματολόγιο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και επομένως ε, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε τον ρόλο αυτό. Μια ερώτηση ή ένα στοιχείο θα ήθελα να αναφέρω. Η αστική ε, πολιτική μας είναι ε, ιδιαίτερος προσφυλής, είναι κάτι πολύ σημαντικό για όλους μας. Η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτά τα πλαίσια ε, είναι ιδιαίτερα ε, ε, σημαντική κατά τη δική μας άποψη. γιατί ξέρετε ότι εμείς είμαστε αυτοί που εκπροσωπούμε τους πολίτες και επομένως και τις διάφορες περιφέρειες ε, προσπαθούμε να βοηθήσουμε ε, και προς εμάς στρέφονται ε, οι πολίτες, όχι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν κάτι δεν πάει καλά. Επομένως θα πρέπει να δούμε το θέμα της συμμετοχής μας, δηλαδή τι, μπορεί, τι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω έτσι ώστε να υπεραμεινθούμε ακόμα περισσότερο των αρχών αυτών. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βαν Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτα απ' όλα, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι σημειώσαμε αισθητή πρόοδο στο θέμα αυτό. Και το σύμφωνο του Άμστερνταμ αρχίζει και λαμβάνει σάρκα και οστά, συγκεκριμενοποιείται αρκετά και ε, μας ενδιαφέρουν αυτοί οι τομείς δράσης που προτείνατε. Συμφωνώ με την κυρία Βέστφαλ. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι νευραλγικός, γιατί τα σχέδια ε, θα έχουν κέρια σημασία για την ε, επίλυση προβλημάτων και εκεί θα πρέπει εμείς ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στους νομοθέτες να διαδραματίσουμε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ερωτώ λοιπόν πώς θα εμπλέξετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτά τα προγράμματα και σχέδια δράσης. Επίσης, ε, πώς βλέπετε τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα προγράμματα που θα, θα χρηματοδοτούνται από τις Καινοτόμε δράσεις ε, από το αστικό θεματολόγιο και πώς ε, θα συνδυαστούν αυτά ώστε να αντλήσουμε τα καλύτερα διδάγματα, πώς θα ενταχθούν στα σχέδια και προγράμματα δράση. Κύριε Μάλετιτς, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρουσίαση. Θα ήθελα να τονίσω ότι είμαι πανευτυχής που τονίσατε πως η γνώση είναι πολύ σημαντική σε αυτά τα σχέδια δράσης, σε την ανταλλαγή εμπειριών και την αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών. Αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε, γιατί όταν έρχομαι σε επαφή με δημάρχους από διάφορα κράτη-μέλη, μου λένε ότι θα ήθελαν κάποιο οδηγό σε επίπεδο πόλων και μάλιστα είναι οδηγό που θα έχει εκπονηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αστική ανάπτυξη και κυρίως τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη που θα είναι και ευφυής, που θα εξορροπεί τις διάφορες διαδικασίες ώστε να καταλήγει στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Αυτό είναι το ζητούμενο, το κοινό σημείο και η κοινή έκκληση των δημάρχων. Επίσης, ε, να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία και για την επιλογή των ε, ε, πρωτευουσών, των ευρωπαϊκών πρωτευουσών, γιατί έχουμε διαφορετικά βραβεία για τις πόλεις. Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα για την επιστήμη, τον αθλητισμό, τώρα έχουμε το καινούριο για την καινοτομία και βραβεία που έχουν κερδίσει η Βαρκελόνη και το Άμστερνταμ. Και όταν ε, ε, βλέπουμε τι μπορεί να γίνει σε επίπεδο πόλης ώστε να κερδιθεί αυτή, αυτό το βραβείο, τότε καλό θα ήταν να εκφωνήσουμε έναν οδηγό, ένα εγχειρίδιο για το τι πρέπει να κάνει μια πόλη για να γίνει πόλη της καινοτομίας και να διεκδικήσει αυτό το βραβείο. Επίσης, οι προτεραιότητες αυτές που αναφέρονται στο σύμφωνο του Άμστερνταμ περιλαμβάνουν και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξη ε, δεξιοτήτων στην οικονομία. Αυτό λοιπόν θα μπορούσαμε να το διασυνδέσουμε με τα σχέδια δράσης και να προτείνουμε έναν οδηγό, ένα εγχειρίδιο για το τι πρέπει να γίνει προκειμένου να διεκδικηθούν τα διάφορα βραβεία σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν αυτό ο οδηγό το χειρίδιο να περιλαμβάνει συγκεκριμένε πληροφορίε για τα βήματα και τι διαδικασίε που θα πρέπει να ακολουθήσει κανεί για να διεκδικήσει ένα τέτοιο βραβείο. Ε, ε, ένα θέμα συναφέ με το προηγούμενο σημείο που εξετάσαμε, την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων. Σε αυτέ τι 12 προτεραιότητε, δεν βλέπω τι δημογραφικέ αλλαγέ, μεν, αλλά μπορούμε να συνδέσουμε μερικέ από αυτές τις προτεραιότητες με τον προβληματισμό των δημογραφικών αλλαγών. Η φτώχεια, για παράδειγμα, η στέγαση, η δημιουργία θέσεων απασχόληση είναι θέματα που συνδέονται και με τι δημογραφικέ προκλήσει. Οπότε πιστεύω ότι και ελπίζω και στο σχέδιο στα σχέδια δράση να βρούμε τη στενή αυτή συνάφεια των προτεραιοτήτων με τις δημογραφικές προκλήσεις. Ευχαριστώ κύριε Μάλετης, ο κύριος Σίσο, Βαλκάρσελ Σίσο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι αν πρέπει να δώσουμε μια επίγουσα άμεση απάντηση στο τι σημαίνει η πολιτική συνοχής, νομίζω ότι θα συμφωνούσαμε όλοι λέγοντας ότι είναι ακριβώς η πολιτική η οποία ε, ε, προσπαθεί ε, ε, να μειώσει τη διαφορά ανάμεσα στις πιο πλούσιες και τις λιγότερο πλούσιες ε, περιφέρειες. Και βεβαίως είναι αυτή η οποία προσπαθεί να δώσει λύση στις κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις. Το θέμα των τοπικών, της τοπικής αντιμετώπισης των προβλημάτων συμπεριλαμβανομένων και της κοινωνικής συμπερίληψης φαίνεται ότι μέσα από τα αστικά θεματολόγια μπορεί ε, να δώσει μια απάντηση ε, και ε, μέσω της αριστείας μπορούμε να προωθήσουμε την, το αστικό θεματολόγιο. Θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στις περιφέρειές μας να αναπτυχθούν στο μέγιστο βαθμό και βεβαίως με τον τρόπο αυτό να μπορέσει και η ύπεθρος να προχωρήσει. Θα πρέπει να ενδυναμωθούν πούμε τα δίκτυα που συνδέουν συνδέουν τις Μητροπολιτικές Αστικές Περιοχές ε, με την ε, Ήπεθρο και δίνουν την ε, δυνατότητα σε όλους να έχουν δυνατότητα πρόσβαση στο χώρο εργασίας. Επίσης η δημιουργία απασχόλησης, θέσεων απασχόλησης είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και φυσικά δεν πρέπει να λησμονούμε σε όλη τη διαδικασία αυτή να διασφαλίσουμε την ισότητα των φύλων. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να σας πω ότι με μεγάλη ικανοποίηση βλέπω την διαδραστική ε, σελίδα του αστικού θεματολογίου ε, αλλά θα πρέπει να μεταφραστεί γιατί τα στοιχεία βρίσκονται μόνο στα αγγλικά και επομένως ε, δεν νομίζω ότι έχουν όλη τη δυνατότητα να τη διαβάσουν. Αν θέλουμε πραγματικά να ενισχύσουμε τη διαδικασία θα πρέπει όλοι να έχουν την δυνατότητα να διαβάσουν όλες τις δυνατότητες που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση Ένωση στη γλώσσα τους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άλμπρεχτ. Ευχαριστώ πολύ. Ήρθα αργοπορημένος γιατί ήμουν ε, στον, ε, στην Επιτροπή Προπολογισμών αλλά ε, γνωρίζω το θέμα και με ενδιαφέρει. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να υπογραμμίσω ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα ο συντονισμός ανάμεσα από τις διάφορες γενικές μεταξύ των διαφόρων γενικών διευθύνσεων και ελπίζω ότι θα υπάρξει επιπλέον συνεργασία και συντονισμό στο μέλλον και μάλιστα όπως είπε και η Ιβάνα προηγουμένως έχουμε μεγάλες ε, ε, έχουμε ε, δραστηριότητες οι οποίες αφορούν την Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης. Υπάρχουν άλλες προτεραιότητες οι οποίες όμως είναι σε άλλη Γενική Διεύθυνση. Εν πάση περιπτώσει εμείς στον Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντα ζητούμε να μην υπάρχουν επικαλύψεις και να υπάρχει περισσότερο συντονισμός. Πάντως είναι θετικό και από εκεί προκύπτει το ερώτημά μου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να χρησιμοποιήσει στο άρθρο 7 ε, για την ε, ε, υποστήριξη των βιώσιμων δραστηριοτήτων με 5%. Εμείς είχαμε ζητήσει και 10% στους επόμενους μήνες να κάνουμε και τη συζήτηση για τη νέα πολιτική συνοχή. Είναι δυνατόν να ενισχυθεί η πολιτική αυτή. Είσαστε διατεθειμένοι να το κάνετε όσον αφορά στην εργασία με το Κοινοβούλιο. Βεβαίω αυτό μας ενδιαφέρει μας πάρα πολύ. Οι συντονιστές νομίζω το έχουν συζητήσει ήδη το θέμα. Είναι σαφές λοιπόν ότι το Κοινοβούλιο θέλει να συμμετάσχει. Όσον αφορά τις εταιρικέ σχέσεις, partnerships, ε, εδώ μεταξύ των ε, ε, μελών ας πούμε συζητούμε τον πραγματικό στόχο των εταιρικών σχέσεων που προκύπτουν, που απορρέουν από το σύμφωνο του Άμστερνταμ. Ποιο είναι το σχέδιο δράση όμως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι περιμένει από αυτές τις 12 ε, ε, ήδη υφιστάμενες εταιρικέ σχέσεις, τι περιμένει από το σχέδιο δράσης. Ε, πρέπει να περιμένουμε κάποιες απόλυτα καινούριε ιδέες, πειραματικές, κάτι απόλυτα καινούριο που δεν θα έχει καμία σχέση με τα όσα υφίστανται ήδη. Ή περιμένουμε, τι περιμένουμε ακριβώς, περιμένουμε να δούμε τρόπους βελτίωσης, διόρθωσης λαθών, ε, τι θέλουμε και από το αστικό θεματολόγιο, καλύτερη νομοθέτηση, απλούστευση της νομοθέτησης, ε, ε, αυτό το σχέδιο δράσης θα έχει κάποιες απόλυτα καινούργιες ιδέες ή θα περιέχει στοιχεία που θα διορθώνουν την υφιστάμενη κατάσταση. Γιατί ξέρετε ότι για τις εταιρικές σχέσεις ε, ε, το θεματολόγιο ξεκινάει από το 17 ε, αλλά τότε 17, 18, 19 δηλαδή αλλά τότε θα πρέπει το νομοθετικό πλαίσιο να είναι ήδη έτοιμο επομένως ερωτώ το νέο σχέδιο δράσης θα είναι ε, εργαλείο για το νέο κανονισμό ή θα είναι παράλληλο με τη διαδικασία του κανονισμού. Δεν είναι ακριβώς ρητορική η ερώτηση, γιατί αν κάνουμε κάτι, το κάνουμε για να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Θεωρούμε λοιπόν ότι ε, το, τα αποτελέσματα ε, που τα διδάγματα των εταιρικών ε, συνεργασιών θα πρέπει να τροφοδοτήσουν την συζήτηση για τον κανονισμό, κατά την άποψή μας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσατε σχόλια, ακούσατε ερωτήσεις. Σας δίνω λοιπόν τον λόγο έτσι ώστε να απαντήσετε στα σχόλια και στις ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ για τις ερωτήσεις, ευχαριστώ για τα σχόλια που είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα. Δεν επεκτάθηκα στη σύντομη παρουσίασή μου σε όλα, αλλά μπορώ τώρα να πω ίσως κάποια παραπάνω πράγματα. Φυσικά και η γνώση είναι θέμα κλειδί, ιδίω γιατί είναι τόσο διαφορετικέ μεταξύ του ε, οι πόλει και σε ό,τι αφορά την πρώτη προκήρυξη, είδαμε με τη γεωγραφική αυτή ισορροπία που θέλαμε να επιδιώξουμε πόσο μικρό κομμάτι καλύψαμε τελικά. Και δυνάμει το άρθρο 7 από το που θέλουμε να εφαρμόσουμε μαζί με τα κράτη-μέλη, μιλάμε για, την υπάρχει αυτή κοινή διαχείριση. Ε, έχουμε κάποιε διατάξει που θα μα βοηθήσουν, έχουμε το δίκτυο ε, και ακούμε τις πόλεις, προσπαθούμε να τις βοηθήσουμε στοχευμένα, ακούγοντας τα προβλήματα και προσπαθούμε να έχουμε στον ατόμο μεγαλύτερη απλούστευση στην ε, πρόσβαση χρηματοδότηση. Αλλά είπα είναι η συνδιαχείριση το θέμα. Ε, τώρα, στην Επιτροπή, τη Δικούσα Επιτροπή, το Steering Committee, χθε είχαμε μια συζήτηση, είχαμε και εργαστήρια σε χώρες της Ευρώπης που δεν είχαμε επιτυχία παρά τις καλές ιδέες, δεν υπήρξε ποιότητα. Ή ανάποδα να υπάρχουν ποιοτικά έργα χωρί καινοτομία. Τώρα όμω βλέπουμε να υπάρχει δυναμικό, να υπάρχουν δυνατότητες, να κάνουμε ό,τι μπορούμε στοχευμένα. Ήμασταν και στη Βουδαπέστη, τη Βαρσοβία, θα πούμε στην Ελλάδα και σε άλλες πόλεις ε, που έχουν το δυναμικό αλλά δεν έχουν ακόμη ε, πετύχει τους στόχους. Ε, αριστεία είναι όρος του 2020, δεν θέλω να συζητήσω για αριστεία, αλλά η υπόθεσή μα είναι ότι αυτή η έννοια τη εφηβεία εξειδίκευση που αφορά και τις πόλει θα οδηγήσει, ε, θα φτιάξει αυτό το διάδρομο που θα οδηγήσει στην αριστεία. Έχουμε και την ανακοίνωση στο Ελσίνκι, τη μεγάλη εκδήλωση για την εφή εξειδίκευση. Θέλουμε υποστήριξη, ώστε και αυτοί που υπολείπονται να κάνουν κάτι. Και ακριβώς η εφής εξειδικεύση είναι η απάντηση. Ξεκινάς με αυτό που έχεις στις περιφέρειες και πάνω σε αυτό οικοδομής και σε κάποια στιγμή στην αριστεία για να μπορεί να ανταγωνιστεί με του υπολείπου σε άλλα προγράμματα. Για τι καινοτόμε δράσει, λοιπόν έχουν στοχευμένη βοήθεια, σκεπτόμαστε πόλεις, βλέπουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη συμμετοχή από όλη την Ευρώπη. Και φυσικά όλα αυτά σε άμεση σχέση με το αστικό θεματολόγιο. Μετανάστευση, σας είπα ήδη ήταν ο στόχος μας, η κινητικότητα. Επιλέγουμε και βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε με βάση αυτό το Και χθε το συζητήσαμε και θα προσπαθήσουμε να συνοψίσουμε τα 18 πρώτα έργα τα οποία εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή και μετά έχουμε τη δεύτερη δεσμίδα που θα εγκρίνουμε φέτο. Και στο δυνατόν πιο σύντομα θέλουμε και να μάθουμε αλλά και να κάνουμε προτάσεις στο πλαίσιο της σχεδίου δράσης. Μπορεί να υπάρχουν κάποια κενά. Θα μπορούσαμε να δείξουμε πώς μπορούν να καλυφθούν τα κενά με ένα καλό project με τους εταίρους μας έχουμε συμφωνήσει να χρησιμοποιήσουμε και τα δίκτυά μας αλλά και ευρύτερα. Κάτι πολύ σημαντικό είναι η φυσικά συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ήταν δεδομένη από την αρχή βέβαια. Τα σχέδια δράσης θα δημοσιοποιηθούν τον Ιούλιο. Και ακόμη και οι όσοι δεν είναι άμεσα ενδιαφερόμενοι καλούνται να πούν ό,τι θέλουν. Βέβαια το σημαντικότερο είναι τώρα, γιατί θα έχουμε τους πρώτους τέσσερις τον Ιούλιο. Αυτό γράφω στην ατζέντα μου, Ιούλιο-Αύγουστο. Τα πρώτα σχέδια δράσης θα είναι έτοιμα τότε. Και βέβαια πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, να έχουμε καλύτερη ομοθεσία. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καθίστεται σαφές ότι θα πρέπει να δώσουμε σημασία στην εδαφική προσέγγιση και η γάμα δελτα άγκρη. Σας δείχνω ότι δεν δουλεύουμε σε στεγανά. Είχαμε το, θεματικό, το θεματολόγιο και για τις αγροτικές περιοχές και συνεργαζόμαστε αυτές οι γενικές διευθύνσεις επειδή υπάρχει αλληλεξάρτηση. Άρα η λειτουργική εδαφική περιοχή είναι η έννοια του μέλλοντος. Στη Γερμανία έχουμε ήδη πολύ μεγάλη πρόοδο. Αυτή λοιπόν είναι η απάντηση και θα πρέπει να το στηρίξουμε και εμείς με τα μέσα μας και στο μέλλον. Την συνεργασία επίσης. Δεν είναι μυστικό. Στην Ευρώπη έχουμε πόλεις ε, μικρής και μεσαίας κλίμακας και έχουμε δύο μετροπολικές μόνο περιοχές στην Ευρώπη. Θέλουμε να στηρίξουμε τη δημιουργία τέτοιων ε, λειτουργικών εδαφικών περιοχών. Υπάρχουν μελέτες και το πρόγραμμά μας είναι μια εξαιρετική μελέτη αυτής της πολυκεντρικής ανάπτυξης. Και σε περιοχές που έχουμε συγκεκριμένες γεωγραφικές ανισορροπίες μπορούμε με τη δική σας υποστήριξη να πετύχουμε πράγματα. Και για το μέλλον. Για το μέλλον, ιδίως για τα ποσοστά, δεν μπορώ να πω πολλά. Uh, αυτό που ε, κάνουμε και τώρα δείχνει ότι υπάρχουν στοιχεία και αυτό θα πρέπει να είναι μία βάση σοβαρή για να εξετάσουμε και αυτό το σκέλος ως ένα μελλοντικό σκέλος πολιτικής. Βέβαια, είναι μια μεγάλη διαδικασία, όπως καταλαβαίνετε. Εμείς θα δώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαρίστω να έρθουμε εδώ να σα τα πούμε όλα. Τα ETIs είναι γύρω στα 200. Αν δεν κάνω λάθο. Και τα μισά μόνο για το αστικό το επίπεδο. Και τα άλλα μισά ε, εδαφικές, ε, λειτουργικές εδαφικές περιοχές. Άρα πηγαίνουμε πολύ καλά, είναι πολύ ενθαρρυντικά τα δείγματα. Αυτή η ταφική προσέγγιση προσλαμβάνει μεγάλη σημασία στις μέρες μας. Έχουμε άλλωστε και τους μεγάλους στόχους της Ένωσης που πρέπει να επιτελέσουν, να επιτύχουμε. Ψηφιακοί στόχοι, ενεργειακοί, μεγάλες προτεραιότητες. Και φυσικά δεν πρέπει να τις διασυνδέσουμε, να υπάρξει αλληλεπίδραση για την επίτευξη των στόχων αυτών. Έχουμε ξεφολογήσει τι εργασίε με τι άλλε γενικέ διευθύνσει. RTD, τι κάνει το ορίζον 2020, τι γίνεται με τι καινοτόμε ενέργειε, γιατί είναι διαφορετικά τα διάφορα εργαλεία. Εμεί κοιτάμε το στο ο Ρίζον κοιτάει πιο πολύ τα θέματα αριστεία. Εμεί προσπαθούμε να δούμε πώ μπορούμε να τα συνδυάσουμε όλα αυτά. Να χρησιμοποιήσουμε καινοτόμε λύσει για να λύσουμε συγκεκριμένα προβλήματα, να τα εξολογήσουμε και να έχουμε μετά οριζόντια κατανομή. Αλλά και άλλα εργαλεία που έχουμε και σε τακτικές συναντήσεις μας ε, ενεργά εργαζόμαστε. Σε ό,τι αφορά τη συμβουλευτική πλευρά, υπάρχει στο σελίδα, όπου αναρτούμε τα πάντα και παρέχουμε στοχευμένες συμβουλές. Έχουμε το focus group και από που να νομίζω ολοκληρώνουμε τις προτάσεις με εσωτερικό επίπεδο, σε επίπεδο πολιτικών γραφείων, τη συμβουλευτική αυτή μια θηρίδα. Θα υπάρχει ένας οδηγός για τις πόλεις και ελπίζω ότι οι πόλεις θα μπορούν να συμβουλευθούν αυτό το δικτυακό τόπο. Αν έχουν πρόβλημα μπορούμε να τους καθοδηγούμε όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν, αλλά και στο πώς θα βρουν τη χρηματοδότηση την αναγκαία. Αυτά έχουμε προβλέψει. Αυτή είναι η στόχη. Ελπίζω να έχω απαντήσει όλες τις ερωτήσεις. Να ξέρετε ότι το αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλη σοβαρότητα το θέμα και στο μέλλον η Επιτροπή σας μπορεί να μας καθοδηγήσει. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you very much. This is for... Σας ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα, οπωσδήποτε θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς αυτή τη διαδικασία του αστικού θεματολογίου και θα έχουμε την ευκαιρία μέσω διάφορων εκδηλώσεων και ε, συναντήσεων να, ανταλλάσσουμε τακτικά απόψεις. Σας ευχαριστώ πάντως που ήρθατε γιατί θα είναι ε, πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και στο μέλλον και θα σας ξανά έχουμε στην Επιτροπή. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που προβλέπει ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το Brexit και την πολιτική συνοχής. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι είχαμε πολλές ε, ευκαιρίες όπου συζητήσαμε το κατά πόσο είναι σκόπιμο να ξεκινήσουμε συζήτηση περί Brexit και Πολιτική συνοχής. Πάντως ε, ακολουθούμε το βασικό σχέδιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως εγκρίθηκε από τη διάσκεψη των Προέδρων και ορίς και πόρισε τον κύριο Φερχόφσα, το συντονιστή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις διαπραγματεύσεις ε, του Brexit, της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ε, ε, η διάσκεψη των Προέδρων ε, ενέκρινε τρία επίπεδα συζήτησης. Στο πρώτο επίπεδο έχουμε τη φάση μέχρι την ενεργοποίηση του άρθρου 50, οπότε διασφαλίζεται μία παρακολούθηση σε επίπεδο διάσκεψη των Προέδρων και εξετάζονται οι συνέπειες του Brexit στις διάφορες πολιτικές που αφορούν τι ε, επιμέρου κοινοβουλευτικέ επιτροπές. Μάλιστα η γραμματεία μας εκπώνησε ένα έγγραφο που το υπέβαλε στου συντονιστές των πολιτικών ομάδων και αυτό είναι ένα ε, τμήμα της διαδικασίας που ακολουθούν και οι υπόλοιπε κοινοβουλευτικέ επιτροπές. Στη δεύτερη φάση, μετά την έναρξη των ε, διαπραγματεύσεων από τη στιγμή που κινητοποιήθηκε δηλαδή το άρθρο 50. Ο κύριος Φερχόφστατ ε, συντονίζει το έργο σε επίπεδο διάσκεψη Προέδρων. Από κοινού με την κυρία Χιούμπνερ που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων καθώς και έχει συντονισμό και με τις ε, επιμέρους επιτροπές για να εξασφαλίσει την εμπειρογνωμοσύνη τους. Στη τελευταία συνεδρίαση της, επισκε... της διάσκεψης Πρόεδρων Επιτροπών, ο κύριος Φερχόφστατ ε, ενημέρωσε το Κοινοβούλιο ότι μετά το πρώτο ψήφισμα που εγκρίναμε στην τελευταία ολομέλεια του Στρασβούργου, πρόκειται να εκπονήσουμε και επιμέρους ε, ψηφίσματα για τομέακες πολιτικές ε, συμπεριλαμβανομένες και τις περιφερειακές πολιτικές. Οπότε θα πρέπει και εμείς να είμαστε έτοιμοι και να έχουμε διαμορφώσει τη θέση της ε, Επιτροπής μας ε, για τα θέματα που μας ενδιαφέρουν κατά την περίοδο των διαπραγματεύσεων. Και στην τρίτη φάση, μετά το πέρας των διαπραγματεύσεων, η Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια με βάση τον ιστορικό κανονισμό για τη διαδικασία συνένεσης, ε, αλλά και οι άλλες συναρμόδιες επιτροπές, θα πρωτοστατήσουν στη διαδικασία. Είχαμε αρκετέ ε, συναντήσεις μέχρι στιγμή στο επίπεδο διάσκεψης πρόεδρων επιτροπών ε, με τον κύριο Φερχόφστατ και τον, και τον κύριο Μπαρνιέ που είναι ε, ο επικεφαλής της ομάδας διαπραγμάτευσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχουμε ήδη εγκρίνει και το πρώτο, πρώτο μας ψήφισμα επί του Brexit. Οπότε σας προτείνω τώρα να ξεκινήσουμε το διάλογο, την ανταλλαγή απόψεων για το Brexit και την πολιτική συνοχής. Θα πρέπει λοιπόν με την ανταλλαγή αυτή απόψεων να προσανατολίσουμε το έργο μας εν ώψη και του ειδικού ψηφίσματος για την πολιτική συνοχής που θα εγκριθεί αργότερα. Εκεί θα πρέπει να αποκρισταλώσουμε τη θέση μας και να δούμε πώς θα συμμετέχουμε στις διαπραγματεύσεις του Brexit για θέματα που φορούν την πολιτική συνοχή. Είδου λοιπόν, περιμένω τις προτάσεις ε, και τα σχόλιά σας. Ο κύριος Όλμπριχτ. Σας ευχαριστώ. Ε, πολλές θα είναι οι συνέπειες του Brexit στην πολιτική συνοχή ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έχουμε άμεσες αλλά και έμεσες συνέπειες του Brexit. Θα πρέπει να δούμε πρώτα ποιες θα είναι οι συνέπειες του Brexit στην πολιτική συνοχή από το 2019-2020 αλλά και μετά. Γιατί αν η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου αποφασίσει να παραμείνει στα προγράμματα της πολιτικής συνοχής Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ε, είναι παρόν στην πολιτική συνοχής μέχρι το 2020 ε, και θα συμμετοχή που θα έχει συνέπειες μέχρι και το 2023. Οπότε είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε τους δημοσιονομικούς πόρους ε, για να ε, βαστιμίσουμε τις υποχρεώσεις μας, γιατί αναφέρθηκαν τα 60 δισεκατομμύρια ανάληψη υποχρεώσεων στην πολιτική συνοχή. Και αυτές είναι οι άμεσες συνέπειες του Brexit για τη συνοχή. Ανακύπτει όμως και το θέμα πώς θα συμμετέχει το Brexit οικονομικά στην πολιτική συνοχή μετά την έξοδό του, δηλαδή μετά το 19 έως το 2023. Βέβαια, έχουμε και κάποιες ήδη ενηλυμένες υποχρεώσεις ε, που θα πρέπει να ε, γίνουν σεβαστές από την Βρετανική κυβέρνηση. Επίσης, αν κρατήσουμε την ίδια μεθοδολογία ε, που είχαμε μέχρι σήμερα, κάτι που δεν είναι σίγουρο, αν θα παραμείνει όμως η μεθοδολογία, 75% του ΑΕΠ, του, του μέσου ΑΕΠ, έχουμε στο ΝΑΤΣ 2. Και δίστανται οι απόψεις. Ποιες θα είναι οι συνέπειες για το μέσο ε, ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τον Brexit. Θα έχουμε αλλαγή του μέσου όρου. Θα μειωθεί ο μέσο όρο του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αν μειωθεί αυτό το μέσο ΑΕΠ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό σημαίνει ότι μερικέ περιφέρειε θα περάσουν από τι λιγότερο αναπτυγμένες στι στις μεταβατικές. Οπότε θα πρέπει να δούμε σε περίπτωση διατήρηση τη μεθοδολογίας ποιε θα είναι οι συνέπειε του Brexit στην πολιτική συνοχή και στο χαρακτηρισμό ενδεχομένω ε, κάποιων περιφερειών ω προ τον ΝΑΤΣ 2 Ή, ίσως θα πρέπει να να αναθεωρήσουμε κάποια κριτήρια της πολιτικής συνοχής, να διαβρύνουμε τα κριτήρια ώστε να μην περιοριζόμαστε μόνο στο ΕΠ, αλλά να έχουμε και άλλους δείκτες της πολιτικής συνοχής. Ίσως θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε και το επίπεδο συγκέντρωση των δεδομένων από το ΝΑΤΣ 2 στο ΝΑΤΣ 3 ενδεχομένω, ε, ώστε να περιλάβει και τα αστικά θέματα. Οπότε δεν θα πρέπει να περιοριστούμε μόνο στην συζήτηση του Brexit, αλλά τη συζήτηση των συνεπειών του Brexit στη δική μας πολιτική και τις πιθανές λύσεις για την επόμενη φάση της πολιτικής. Και υπάρχουν και άλλα στοιχεία, αλλά δεν έχουν άμεσο σύνδεσμο με το Brexit. Αλλά είναι σημαντικά για την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Διερωτώ με λοιπόν ποιες θα είναι οι συνέπειες στην πολιτική συνοχή μιας Ευρώπης δύο ταχυτήτων. Η πρόταση για τον προπολογισμό της, ε, της δημοσιονομικής ικανότητας Ευρωζώνης. Και αυτή θα είναι μία από τις συνέπειες του Brexit. Γιατί είναι ακόμη ανοιχτή η συζήτηση αν θα έχουμε προπολογισμό τη Ευρωζώνη. Γιατί αν θεσπιστεί προπολογισμό τη ε, Ευρωζώνη, ποιε θα είναι οι συνέπειε του στην πολιτική συνοχή. Αυτό δεν είναι άμεση συνέπεια, αλλά έμεση συνέπεια του Brexit. Επίση, ε, τι θα γίνει για την περίοδο 2014-2020 και τι γίνεται για την περίοδο μετά το 2020 σε ό,τι αφορά τι συνέπειε του Brexit. Σα ευχαριστούμε. Ο κύριος Μποστινάρου, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ακολουθήσω την ε, γραμμή σκέψης του Γιάννου. Γιατί υπάρχουν ε, πολλαπλά επίπεδα ε, μέσω των οποίων θα επηρεαστεί η περιφερειακή πολιτική από το Brexit. Το θέμα είναι πώς να αξιολογήσουμε σωστά εκ των προτέρων τον αντίκτυπο αυτό έτσι ώστε να μειώσουμε ε, τι το εύρος των αντικτύπων αυτών. Όλη η διαδικασία αυτή του Brexit, όταν θα έχει φύγει δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει να αξιολογηθεί ποια είναι η κατάσταση συνολική και μετά βεβαίως γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία προσπαθούν να εκμεταλλευτούν ε, το ε, ε, Brexit για να αλλάξουν την πορεία της πολιτικής συνοχής. Ξέρουμε από την επιχειρηματολογία τους για τους λόγους για τους οποίους θέλουν να αλλάξουν την πολιτική συνοχής λόγω του ότι η βάση του ότι εγκαταλείπεται το Ηνωμένο Βασίλειο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτο ερώτημα, ποιες είναι οι επιπτώσεις ε, για τις ε, δύο μεγάλες ομάδες, για τους καθαρούς συνεισφέροντες και τα κράτη συνοχής. Οι καθαροί συνεισφέροντες έχουν την τάση να εκμεταλλευτούν τον, το Brexit ε, έτσι ώστε είτε να μειώσουν τις συνεισφορές για την συνοχή είτε έτσι ώστε να έχουν μια κατά τη δική τους άποψη καλύτερη συμφωνία γνωρίζοντας ότι μερικές φορές ε, ο συμβιβασμός μπορεί να υπονομεύσει το μέλλον της ε, πολιτικής συνοχής ε, και επίσης, πολύ σημαντικό επίσης και να μην το υποτιμούμε, πολύ σημαντικό λέω είναι να δούμε εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μελετά το γεγονός ε, η σκοτή σκοτία ε, να, το ενδεχόμενο μάλλον η σκοτία να παραμείνει ε, στην πολιτική συνοχής. Ε, είναι δύσκολο να απαντηθεί το ερώτημα αυτό, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε στις λεπτομέρειες τους τις διάφορες αποχρώσεις των ερωτημάτων που προκύπτουν από το Brexit σε σχέση με την πολιτική συνοχής και βεβαίως και μαζί με το επίπεδο ΝΑΤΣ 2 και τα υπόλοιπα ε, όλα θα πρέπει να συζητηθούν εντελεχώς πριν ξεκινήσει η μεγάλη συζήτηση στην Επιτροπή μας για το μέλλον της πολιτικής συνοχής και την επίπτωση που θα έχει το ζήτημα στις διάφορες εκθέσεις και τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουν το θέμα οι διάφοροι εισηγητές. Ευχαριστώ κύριε Μποστινάριο, κυρία Μπρέσο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως ανέφεραν ήδη οι συνάδελφοι, αντιμετωπίζουμε δύο προβλήματα. Το ένα είναι σημαντικό, γιατί βεβαίως πρέπει να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η φάση της πολιτικής συνοχής, δηλαδή θα πρέπει να έχουμε βεβαιότητες και όσον αφορά τη συμμετοχή μέχρι το τέλος της περίοδου που δεν είναι το 2020 ε, αλλά το 2023 γιατί υπάρχουν και τα διάφορα συμπληρωματικά στοιχεία Κατά πόσον δηλαδή θα παραμείνει ε, μέχρι το τέλος ε, η η... το Ηνωμένο Βασίλειο, όχι μόνο από οικονομικής πλευράς, αλλά και από άλλων ε, στοιχείων πολύ σημαντικών. Υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα, πολύ σημαντικό πώς θα επαναπροσδιοριστεί η πολιτική συνοχής ε, από τη στιγμή που δεν θα είναι ε, ε, παρούσα δεν θα είναι παρόν το Ηνωμένο Βασίλειο με αυτή την υποσημείωση της Σκοτίας που αναφέρθηκε προηγουμένως. Νομίζω ότι εδώ μιλάμε για μια μεγάλη χώρα ε, η οποία βγαίνει, μια μεγάλη χώρα με υψηλό εισόδημα και επομένως υπάρχουν πολλά ε, ζητήματα τα οποία προκύπτουν ε, και αλλάζουν και οι ισορροπίες ανάμεσα στις άλλες χώρες. Οπωσδήποτε θα είναι πολλές οι περιφέρειες οι οποίες τώρα βρίσκονται ε, στην συνοχή που θα γίνουν πλέον μεταβατικές ε, περιφέρειες. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας υποβάλει κάποιες εκτιμήσεις στοιχείων για το ΑΕΠ, ε, τι θα προκύψει με την τροποποίηση των στοιχείων ΑΕΠ, πώς αλλάζει, ε, η, ε, ε, πώς αλλάζει ο χάρτης της Ευρώπης όσον αφορά τη συνοχή μέσα του ΑΕΠ και τα Ίσως πρέπει να πούμε ότι εμείς μάλλον είμαστε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή η οποία ξεκινάει τη συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Όλοι καλούμεθα να συμμετάσχουμε σε ανταλλαγή απόψεων και σκέψεων ε, με τους εμπλεκόμενους ε, φορείς δημοσίους, ιδιωτικούς κτλ. Και οπωσδήποτε πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε κάποιο προσανατολισμό. Ε, και ε, ακόμα περισσότερο που η νέα κοινωνική πολιτική, ε, η συγγνώμη, πολιτική συνοχής θα ξεκινήσει ήδη από τώρα και όχι μετά την έναρξη της επόμενης θητείας. Τώρα προετοιμάζουμε το 2020. Απ' την άλλη πλευρά δεν έχουμε στη διάθεσή μας τα οικονομικά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα έτσι ώστε να ξεκινήσει η συζήτηση και μεταξύ των χωρών και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βεβαίω, είναι δεδομένο ότι την πολιτική συνοχή θα την υπερασπιστεί η Επιτροπή μας. Δεν είναι δεδομένο ότι θα την υπερασπιστεί το σύνολο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να βασιστούμε σε μια αξιολόγηση σωστή και ρεαλιστική των διαφόρων εναλλακτικών τι σημαίνει για τις διάφορες χώρες η κάθε περίπτωση. Υπάρχουν ε, χώρες ε, ε, οι οποίες είναι καθαροί συμβάλλοντες αλλά αντιμετωπίζουν προβλήματα. Αναφέρομαι στη χώρα μου, σκέφτομαι τη χώρα μου. Ε, έχουμε πολλές χώρες η κατάσταση των προϋπολογισμών και των ισολογισμών των οποίων απαιτεί σοφροσύνη στην ε, διαχείριση ε, και στον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει όλα τα στοιχεία αξιολόγησης έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε πλέον συγκεκριμένες εναλλακτικές λύσεις από τον οποίο να συζητήσουμε. Και βεβαίως το θέμα των ε, συνεισφορών είναι πολύ σημαντικό στα πλαίσια του Brexit. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχουν ε, επιτροπές οι οποίες ε, ενδιαφέρονται ίσως περισσότερο για τα νομικά ζητήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά αλλά εμείς εδώ έχουμε μελήματα και προβληματισμούς που αφορούν τα χρήματα, που αφορούν τη συνοχή και επομένως νομίζω ότι στη δικιά μας Επιτροπή θα πρέπει να έχουμε ένα σαφές πλαίσιο. Μάλλον η Επίτροπος θα πρέπει να μας δώσει ένα σαφές πλαίσιο, γιατί αυτό θα είναι πολύ χρήσιμο για όλους μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νίκολσον έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ξεκαθαρίσω ότι εδώ εκπροσωπώ τον κύριο Λούρ, το συντονιστή από του συντηρητικού. Άρα αυτά που θα σας διαβάσω δεν είναι δικά μου λόγια. Άρα μην πυροβολείτε τον αγγελιαφόρο παρακαλώ. Εγώ απλά μεταφέρω άλλων μηνύματα. Βέβαια, ίσως στο τέλος να κάνω και κάποια δικά μου σχόλια. Το λέω όμως ευθύς εξ αρχής, ε, ότι εκπροσωπώ τον κύριο Λούρ που σας ευχαριστεί πολύ κυρία Πρόεδρε που έχετε συμπεριλάβει στη μέση διάταξη του θέμα αυτό, το Brexit σίγουρα θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στο μέλλον της πολιτικής συνοχής ε, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το Brexit θα επηρεάσει και τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις ε, για την περίοδο την επόμενη, αλλά και το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό. Είτε θα έχουμε μικρότερο προϋπολογισμό συνοχής, είτε περισσότερες ε, υποχρεώσεις μετά το 2020 για τους καθαρούς εισφορείς. Σίγουρα το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνουν φιλόδοξε αλλαγέ στην πολιτική συνοχή ε, και είναι πολύ καλό που γίνεται αυτή η ανταλλαγή απόψεων ε, με υπόβαθρο την έκθεση Westphal που κάνει ένα απολογισμό των διδαγμάτων που αντλήσαμε τον κανονισμό περικοινών διατάξεων και θα τα συζητήσουμε και στο πλαίσιο του ΣΓΑΡΕΚ του επόμενου πολιετούς. Κάποια σχόλια. Η Πρωθυπουργός στο γράμμα, στην επιστολή της ε, στις 29 Μαρτίου προς τον Πρόεδρο Τούσκα μιλά για μια σχέση εταιρική, βαθιά εταιρική σχέση μετά το Brexit. Άρα ακόμα και όταν δεν θα έχει άμεσο ρόλο και άμεση χρηματοδοτική συνδρομή το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν θα είναι αποδέκτης ε, των επενδυτικών και διαφορετικών ε, ταμείων, θα έχει παρόλα αυτά ρόλο και γι' αυτό πιστεύω ότι εξακολουθούν να υπάρχουν τομείς αμπέας συνεργασίας. Πρέπει να διδαχθούμε ένας από τον άλλο. Ε, σε ό,τι αφορά τα διάφορα συστήματα περιφερειακής χρηματοδότηση και θα συνεχίσουμε να ανταλλάσσουμε γνώσει και εμπειρία και σε ακαδημαϊκό και σε πρακτικό επίπεδο. Δεύτερον, όπω λέγεται και στην επιστολή ΣΑΜΕΗ, υπάρχουν κάποιοι τομεί που η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θέλει να έχει οικονομική συνεργασία. Και ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν στους επόμενους μήνες και πρόσφατα το ανέφερα στην Επιτροπή είναι η συμμετοχή της Βρετανία στην ΕΤΕΠ. Η ΕΤΕΠ θα είναι σίγουρα ένα από τα κομβικά θέματα. Βλέποντας όμως το μέγεθος της οικονομικής συνδρομής του Ηνωμένου Βασιλείου στην τράπεζα, θα είναι αμοιβαία αποφελές το να συνεχίσει να συμμετέχει το Ηνωμένο Βασίλειο σε αυτήν την τράπεζα. Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων θα συζητηθούν και από τι δύο πλευρές ε, ζητήματα και υπάρχουν διαπραγματευτά ζητήματα και από τι δύο πλευρέ, όμω θα χρειαστεί να γίνουν υποχωρήσει και από τι δύο πλευρέ. Τρίτον, σε ό,τι αφορά την πολιτική συνοχή, ίσω το πιο λεπτό ζήτημα θα είναι οι οικονομικέ δεσμεύσει τη Βρετανίας και πώς αυτές θα ενταχθούν ε, στο λογαριασμό του Brexit όταν φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο το 2019. Όχι μόνο το 30% των κονδυλίων, όπως ήδη υπόθηκε σήμερα, στο πλαίσιο του πολίτου θα έχουν δαπανηθεί, αλλά θα υπάρχουν και υπάρχουν και νομικά επιχειρήματα που λένε ότι θα πρέπει να συνεχίσει να συμμεσφέρει το ΕΕ και μετά το Brexit. Θα πρέπει αυτέ τι συζητήσεις να τι δούμε με ανοιχτό πνεύμα, Ξέροντα ότι αυτό που επιδιώκει η Ένωση δεν είναι ένα νορβηγικό μοντέλο, αλλά μια σχέση μοναδική με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, για τα επόμενα δύο χρόνια η ομάδα ECR θα συνεχίσει να εργάζεται σκληρά και να μελετά αυτά τα ζητήματα που θεωρούμε ότι είναι σημαντικά για την ε, πολιτική συνοχή. Μείωση γραφειοκρατία και γραφειοκρατικού διοικητικού άχθου, εξορθολογισμό, οικονομικών μέσων, μεγαλύτερη ευελιξία, επενδύσει και επίσης ε, ε, συνετές ε, δημόσιες δαπάνες. Αυτά είναι τα βασικά θέματα. Ο κ. Λούρ θα συνεχίσει να συνεργάζεται και στο πλαίσιο της ΙΑΡ αλλά και στο πλαίσιο αυτής της Επιτροπής με τους συναδέλφους του και αυτές τις προτεραιότητες. Αυτά είναι αυτά που είχε να πει ο κ. Λούρ. Χαίρομαι που διάβασα αυτά που είχε να πει ο κ. Λούρ. Αλλά τώρα, εξ ονόματός μου, και όχι εξ ονόματος του κ. Λούρ, Άκουσα να αναφέρει τη Σκοτία και τι θα γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εγώ πιστεύω βαθιά και ήμουν πολύ καιρό στην πολιτική, πιστεύω στην πολιτική και αν δείτε τι έγινε μέσα σε μια εβδομάδα, έχουμε εκλογέ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Που μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα όπω προχωράμε. Σε ό,τι αφορά τη Σκωτία. Εγώ είμαι από τη Βόρεια Ιρλανδία. Η Βόρεια Ιρλανδία ψήφισε να παραμείνει κι αυτή. Το ενωμένο Βασίλειο όμω προσχώρησε τότε στις κοινότητες ευρωπαϊκές και έτσι θα αποχωρήσουν. Ε, θα αποχωρήσει ως Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο σκότος που μπορεί να μιλήσει για τη σκοτή, γιατί δεν θέλω εγώ να τους ε, εκπροσωπήσω. Αλλά μην περιμένετε, μην κρατήσετε και την αναπνοή σας για το τι μπορεί να γίνει. Ποια είναι τα προβλήματα και στη δική μου την περιοχή, στην Βορειοελλανδία θα είμαστε το μόνο μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου που θα έχει ερσαίο σύνορο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου καθιστά σαφέ, σε μένα τουλάχιστον, αλλά και σε όλους, το είπε και η Πρωθυπουργό, ότι θέλει να είναι ομαλά, να είναι μάλλον ενιαία τα σύνορα ε, και αυτό ζήτησε και αυτό το δέχομαι. Όμως, να πω ότι αν δεν είναι στην ενιαία αγορά στην Τελωνιακή Ένωση του Ενωμένου Βασίλειου. Πώς θα έχει αυτό το ενιαίο σύνολο το ε, σίδερο χωρίς ε, Δεν μπορώ να το καταλάβω. Σκληρά σύνορα μεταξύ Βόρειας Ιρλανδίας και Δημοκρατίας Ιρλανδίας δεν τα δέχομαι και δεν το προτείνουν βέβαια. Όμως δεν θα δεχτώ και σύνορα μεταξύ Βόρειο Ιρλανδίας και λοιπού ε, Ηνωμένου Βασιλείου. Και δεν θέλω να λυθεί ένα πρωινό 4 το πρωί στη Ριντελαλουά σε ένα κτίριο ε, μέσα ε, στην κούραση που θα έχουν όλοι αυτοί οι διαπραγματευτές τότε γιατί είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα αυτό και πρέπει να αντιμετωπιστεί ε, στις διαπραγματεύσεις είναι άκρο σημαντικό για όλους τους Βορειοϊρλανδούς και όχι μόνο για αυτούς για όλους τους Ιρλανδούς που εξαρτώνται από το εμπόριο μεταξύ των δύο αυτών περιοχών. Μίζον το πρόβλημα, λοιπόν, και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και νομίζω ότι η Επιτροπή μας έχει το ρόλο της να διαδραματίσει. Ήμουν συντονιστής ε, ε προσπάθησα να καλύψω τα θέματα του περιβάλλοντος μεταξύ άλλων και το αλίας. Σε πολλά χρόνια έχω εμπειρία. Θα συνεχίσω να προσφέρω τις υπηρεσίες μου, αλλά πρέπει να σας πω ότι πρέπει να παραμείνουμε ευέλικτοι και να μπορούμε να προσαρμοζόμαστε στη ροή των εξελίξεων. Ευχαριστώ μεταφέρετε, θα ήθελα να μεταφέρετε και στον κύριο Λούερ ε, τις ευχαριστίες μας που εξέφρασε τη θέση του μέσω ημών. Η κυρία Μάλετιτς, ε, οι καινοτομίες ε, και οι αβεβαιότητες είναι από τις βασικές προκλήσεις της νέας της περίοδου που διανύουμε, γιατί είχαμε πολλές ναι, πολλά, πολλές πολλά νέα στοιχεία και αυτό μα δημιουργεί πολλέ ε, αβεβαιότητε και απορίε ε, και για τη νέα περίοδο. Γι' αυτό θέλουμε τη βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να ε, διορθώσουμε αυτές τις αβεβαιότητες, να διασκεδάσουμε αυτές τις αφιβολίες για να δούμε τι μέλη ενέστε με βάση διαφορετικά σενάρια, όπως είπε και η κυρία Μπρέσο. Επίσης, θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επόμενη περίοδο να μην προσθέσει νέα στοιχεία και να έχει έτοιμο τον κανονισμό μέχρι το, του 2018, γιατί από το 2019 θα έχουμε τις ε, νέες εκλογές, νέες ευρωεκλογές. Οπότε δεν μπορούμε να περιμένουμε το 2020 για να ε, θεσπίσουμε τα νομοθετικά μέτρα και τα νέα δομικά στοιχεία της ε, πολιτικής συνοχής για τη νέα περίοδο στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει όλα πολύ πιο νωρίς να τα έχουμε καθορίσει. Χθες μιλήσαμε και για τις εκ των προτέρων ερεσιμότητες. Ε, είμαστε ήδη στην τέταρτη χρονιά εφαρμογής ε, και μας δυσαρεστεί το γεγονός ότι πολλές εκ των προτέρων ερεσιμότητες δεν έχουν ακόμη αυτό είναι απαράδεκτο και αυτό συνέβη γιατί δεν είχαμε θεσπίσει αυτές τις των προτέρων αρεσιμότητες αρκετά έγκαιρα. Αυτές θα πρέπει εμπρόθεσμα κατά την έναρξη της περίοδου να προσδιορίζονται οι εκ των προτέρων αρεσιμότητες και όχι στη μέση περίοδου. Θα πρέπει να... Είμαστε έτοιμοι εμπρόθεσμα έγκαιρα πριν την έναρξη περίοδου. δε μη θα έχουμε και πάλι στην επόμενη περίοδο το ίδιο πρόβλημα της ε, ε, μη υλοποίηση των στόχων της πολιτικής συνοχής. Και όλοι θα αρχίσουν να αφισβητούν την ίδια τον ίδιο το λόγο ύπαρξης και την αναγκαιότητα της πολιτικής συνοχής εξαιτίας αυτής της καθυστέρησης και της ολιγορίας. Ευχαριστώ κύριο Σκάρβαρ. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η διαμόρφωση της θέσης της Βρετανικής κυβέρνησης ε, άλλωστε επίκυνται και βουλευτικές εκλογές όσον όπου θα πρέπει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η θέση της νέας κυβέρνησης. Πάντως συμφωνώ ότι θα πρέπει να ξανασκεφτούμε τα κριτήρια, να επαναπροσδιορίσουμε τα κριτήρια της συνοχής, όπως είπε ο κ. Σόλμπριχτ. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως θεσμικό όργανο θα πρέπει να εγκύψει σοβαρά στο θέμα αυτό. Επίσης, δεν ξέρω ποιος μίλησε για την Ευρώπη των δύο ταχυτήτων, και αυτή δεν θα είναι η συνέπεια του Brexit η Ευρώπη δύο ταχυτήτων αλλά τη ύπαρξη Ευρωζώνη ε, και χωρών εκτό Ευρωζώνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ο λόγο ύπαρξη ε, δύο ταχυτήτων. Επίση, ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτά τα θέματα δεν είναι μόνο συνέπειε του Brexit. Και δεν υπάρχουν μόνο. Θα πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι υπάρχουν δύο επιλογές. Είναι, είναι κανείς ε, εντός ή εκτός Ευρώπης. Δεν μπορεί να διαλέγει ότι το συμφέρει. Επίσης, ε, το γεγονό ότι υπάρχει πυρήνες Ευρωζώνης και χώρες που είναι εκτός Ευρωζώνης ήδη de facto δημιουργεί δύο διαφορετικά επίπεδα. Μάλιστα, ε, μερικές αποτυχίες ευρωζώνης ε, οδήγησαν σε μεγάλη ανισότητα ακόμη και εντός ευρωζώνης εξαιτία της ε, δυσχερούς οικονομικής κατάστασης σε χώρες όπως η Πορτογαλία, Ελλάδα, Ιρλανδία και ούτω καθεξής. Και πάλι τον Ιούλιο θα έχουμε τον πονοκέφαλο της Ελλάδας και πολύ πιθανό και μια αθέτηση υποχρεώσεων η πληρωμών. Επίσης, η στάση απέναντι στη Σκοτία και η πιθανότητα παραμονή της Σκωτία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς είμαστε ε, Ηνωμένο Βασίλειο ε, που περιλαμβάνει και τη Σκοτία και την Βόρεια Ιρλανδία και πιστεύουμε ότι και μετά τον Brexit η Ένωση θα γίνει πιο δυνατή. Θα πρέπει να περιμένουμε βέβαια και την έκβαση ε, των εκλογών στην ε, Σκοτία. Θα είναι δύσκολο το αποτέλεσμα και πολλοί ήδη στη Σκοτία ξέρουν ότι έχουν περισσότερα περιμένουν από το Ηνωμένο Βασίλειο από ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε θα πρέπει να δούμε τον διάβολο που κρύβεται στι λεπτομέρειε και μετά το νέο δημοψήφισμα. Πάντω και στη Βόρεια Ιρλανδία και στη Σκωτία, όντω η πλειοψηφία τάχθηκε υπέρ τη παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου. Αλλά το πλαίσιο αλλάζει. Και δεν έχω τα στοιχεία για την Βόρεια Ιρλανδία, αλλά για τη Σκωτία είναι σαφέ ότι έχει αυξηθεί η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εσωτερικό της Σκοτίας. Θα πρέπει πάντως να φερθούμε ως ε, ενήλικες και να το, να το δούμε πολύ όρημα το θέμα αυτό. Πάντως, επειδή έχω και οικογένεια κοντά στα σύνορα, το θέμα του σκληρού σύνορου είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα είναι πρόβλημα για τη Βόρεια Ιρλανδία. Και όλοι μιλούμε για τις ειδικέ σχέσεις μεταξύ της πατρίδας μου και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και εγώ βλέπω ε, όμως ε, ιδιαίτερες σχέσεις ε, με την Ιρλανδία και το, μεταξύ Ιρλανδίας και Ηνωμένου Βασίλειου. Νομίζω ότι αυτό είναι πιο σημαντικό. Και Όσο μάθα πρέπει να δούμε πώς θα αλλάξουν και οι σχέσεις της Ιρλανδίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη στιγμή που θα υλοποιηθεί το Brexit. Γιατί όντως έχουμε ειδικέ σχέσεις, ε, ιδιαίτερες σχέσεις με την δημοκρατία της Ιρλανδίας. Και εγώ ε, θα είμαι κατά, θα ε, κατά του σκληρού συνόρου μεταξύ Βορείου Ιρλανδίας και Ιρλανδίας. Νομίζω ότι κανένας δεν είναι υπέρ ενός σκληρού συνόρου. Εγώ πιστεύω ότι μπορούν να συναυθούν διμερείς συμφωνίες και έχω μεγάλη αισιοδοξία γι' αυτό. Η Ελλαδία ε, ήταν μια πιο, υπέρ μιας πιο ελαστικής προσέγγισης της πολιτικής συνοχής. Αυτά, ευχαριστώ. Thank you. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Όμπριχτ, έχετε το λόγο. Μια μικρή διευκρίνηση, σύντομη διευκρίνηση να, για να πω ότι βεβαίως ε, αυτή η Ευρώπη δύο ταχυτήτων που ανέφερα δεν είναι αποτέλεσμα του Brexit. Δεν το είπα ποτέ αυτό, ούτε το πιστεύω. Ωστόσο, πολλές συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή, συζήτηση, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πάγωσαν τη στιγμή που πήρε την σχετική απόφαση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επομένως, ναι, αυτό που ανέφερα δεν ε, είναι άμεση απόρρια του Brexit, αλλά στην έκθεση Μόντι αναφέρεται καθαρά ότι ε, άνοιξε ένα παράθυρο ευκαιρίας να ξαναανοίξουν ε, συζητήσεις παλιές. Είναι λίγο το, σαν να ανοίξαμε το κουτί της Πανδώρας. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν πράγματα τα οποία πυροδοτήθηκαν από τον Brexit, χωρίς να είναι όμως αν έχουν άμεση σχέση να είναι απόρρια του Brexit όχι επειδή έγινε το Brexit, ε, προέκυψαν τα ζητήματα αυτά, αλλά επειδή είχαν την ευκαιρία να ξανα... Ναι, εντάξει, ε, ε, δεν είπα και εγώ, είπα, να σας πω και κάτι, ότι... Εγώ μιλάω σαν Άγγλος στο Ηνωμένο Βασίλειο και ε, να σας πω ότι στην Αγγλία είναι διαφορετική η άποψη που έχουμε ε, για την, ε, για την περιφερειακή πολιτική και για την πολιτική συνοχή στο θα ας πούμε ή στην Μητροπολιτική Περιφέρεια αυτή έχουμε τελείως διαφορετική άποψη για την περιφερειακή πολιτική την βλέπουμε με πολύ θετικό μάτι ξέρω ότι αλλού την βλέπουν διαφορετικά ε, πρόεδρος. Είμαστε πολύ ανοιχτοί στη συζήτηση στην ε, Επιτροπή μας ε, και δεν θέλουμε βεβαίως να γίνει μια συζήτηση μεταξύ των δυο σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, λέει η Πρόεδρος, για την συμβολή σας σε αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων. Συμφωνώ, συμφωνώ με προλαλήσαντες που είπαν ότι υπάρχουν ε, ζητήματα ε, πολύ σημαντικά τι θα γίνει από το 14 μέχρι το 20 στην περίοδο αυτή, ε, πώς θα ολοκληρωθεί η περίοδος, τι μπορούμε να περιμένουμε όσον αφορά τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου μετά, για τη συμμετοχή του μετά από το 18 ή το 19 όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις του Brexit. Δεύτερον, το θέμα του προϋπολογισμού και ποιος θα είναι ο βαθμός αναδιανομής μεταξύ των κρατών μελών. Θα είναι λιγότερος για όλες τις περιφέρειες ή για ορισμένες από τις περιφέρειες. Αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Αυτά που ακούσαμε ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης ε, είναι σχετικά ερωτήματα. Τρίτον, είναι σημαντικό να δούμε πώς ε, θα αλλάξει η ταξινόμηση των ε, περιφερειών ε, σύμφωνα με την μεθοδολογία που ακολουθούμε τώρα θα προκύψουν σημαντικές αλλαγές όσον αφορά την ταξινόμηση των περιφερειών. Θα πρέπει να το δούμε. Και θα μπορούσα να προσθέσω και κάτι άλλο. Άλλο ένα σημείο, το οποίο σχετίζεται με τα όσα είπε ο κύριος Νίκολσον. Εδώ μιλάμε για εδαφική συνεργασία και ο ρόλος ε, του Ηνωμένου Βασιλείου σε κάποια υπερθνικά ε, κυβερνητικά προγράμματα ε, είναι πολύ σημαντικός όχι μόνο για το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά για άλλες γειτονικές χώρες στην προκείμενη περίπτωση το θέμα με της Βόρειας Ιρλανδίας και της ειρνευτικής διαδικασίας στη Βόρεια Ιρλανδία αποτελεί ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Δέχομαι την πρότασή σας να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιο λεπτομερείς πληροφορίες. Θα το, θα το διευθετήσουμε με την γραμματεία έτσι ώστε να προετοιμαστούμε καλύτερα στις μελλοντικέ συζητήσεις και να προετοιμάσουμε καλύτερα τη θέση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης στις μελλοντικέ συζητήσεις. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την ε, συζήτηση που είχαμε. Ολοκληρώσαμε λοιπόν ε, με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Το επόμενο θέμα προβλέπει την έγκριση των αποφάσεων των συντονιστών. Ε, οι συντονιστές συναντήθηκαν, συνεδρίασαν χτες και δόθη και σας εστάλει χθε το βράδυ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το σύνολο των αποφάσεων των συντονιστών μπορούμε να τις υπερψηφίσουμε. Ναι, τεκμέρο διότι δεν ακούω παρατηρήσεις. Υπό τα διάφορα έχετε κάτι, θέλετε να σημειώσετε κάτι υπό τα διάφορα. Όχι από ό,τι βλέπω. Να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε έκτακτη συνεδρίαση στο Στρασβούργο της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης την 18η Μαΐου από τις 11 μέχρι τις 12 το πρωί. Αυτή θα είναι η επόμενη συνεδρίασή μας. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, τους διερμηνείς, λέει η Πρόεδρος, που μας βοήθησαν στη διάρκεια της συνεδρίασή μας ε, και κλείνει η συνεδρίαση της Επιτροπής.